Not uh, Συνάδελφοι, θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχετε εξετάσει την ημερήσια διάταξη. Εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρείται δεκτή. Να χαιρετήσω εδώ τους εκλεκτούς εκπροσώπους και της Λιθουανικής Προεδρίας, την οποία χαιρετίζω χωρίς να βλέπω όμως, δεν ξέρω που είναι, κάπου θα είναι πάντως. Α, στη θέση της πάντα. Voilà. Et je salue Χαιρετίζω επίσης και τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος και αυτός κάπου στην αίθουσα είναι. Με πουκαμισάκι βλέπω κύριε Διευθυντά. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του πήραν το σακάκι μάλλον. Λοιπόν, είμαστε στην αίθουσα η οποία ονομάζεται αίθουσα συνδιαλλαγής. Κάτι το οποίο δεν είναι και ιδανικό για τις εργασίες μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Αλλά μιας και απλά θα προσπαθήσουμε να δούμε τις, ε, την κατάληξη των διαπραγματεύσεων των δημοσιονομικών, νομίζω είναι ευνοϊκό το κλίμα. Χαιρετώ επίσης τους, ε, τους ε, επισκέπτες. Θα έχουμε μια σημαντική αντιπροσωπή από την Πορτογαλική τηλεόραση, η οποία ακόμα δεν έχει φτάσει και θα τους χαιρετήσουμε όταν φτάσουν διότι κάνουν ένα ρεπορτάζ για τους Πορτογάλους Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εξάλλου, στα πλαίσια των ανακαινώσεων του Προέδρου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας την Κοινοβουλευτική Εβδομάδα του έτους 2014 που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου ήδη του 2014. Γιατί αυτό, ξέρετε ότι για τρία συνεχή ετή οργανώσαμε στην αρχή του χρόνου διακοινοβουλευτικές συναντήσεις με τους ομολόγους μας από τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Εδώ και δύο χρόνια οι συναντήσεις αυτές πήραν τη θέση τους επίσημα στα πλαίσια της λεγόμενης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τη στιγμή κατά την οποία παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Αιτήσει προοπτικές ανάπτυξης και το Συμβούλιο Κορυφής του μηνός Μαρτίου, το οποίο καθορίζει τις πρώτες προτεραιότητες για την οικονομική πολιτική των κρατών μελών. Ανάμεσα στις δύο αυτές συναντήσεις εκφράζονται και τα κοινοβούλια. Φέτος η διάσκεψη προβλέπεται λοιπόν στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου και θα έχει πάρα πολύ μεγάλη νομίζω σημασία γιατί την ίδια εβδομάδα και για ένα τριήμερο θα ε, συνέλθει η διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία η οποία όπως είπα έχει πλέον έναν διοργανικό επίσημο θα έλεγε κανείς χαρακτήρα και από την άλλη η διακοινοβουλευτική συνάντηση που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Fiscal Compact. όπου ε, συνεδριάζουν από κοινού εκπρόσωποι των κρατών μελών, των κοινοβουλίων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 25 από 28 χώρες που συνεδρίασαν στο Βίλνιους πριν ένα μήνα και θα συναντηθούν ε, την, στην επόμενη συνάντησή τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής της διακοινοβουλευτικής. Αυτό γίνεται εδώ λοιπόν στις Βρυξέλλες και θα σας το ξαναθυμίσω βέβαια μέχρι τότε, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι ευρωβουλευτές μας να είναι παρόντες ιδιαίτερα στην απογευματινή συνεδρίαση, σε μία απογευματινή, η οποία θα είναι συνάντηση αποκλειστικά ανάμεσα στους συναδέλφους των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών και στα μέλη μας. Θα συναντηθούν και με την Επιτροπή ΕΚΟΝ και με την Επιτροπή Απασχόλησης, που και αυτοί οργανώνουν συναντήσεις, αλλά θα έχουμε μια ειδική συνάντηση λοιπόν εδώ εμείς με τους συναδέλφους, τους εθνικούς συναδέλφους, και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, την αντιπροσωπεία μας σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. Η ποιότητα φυσικά θα δοθεί από τους Πορτογάλους συναδέλφους και η ποσότητα από όλους τους υπολείπους. Τα λέω αυτά αστεία για την ε, πορτογαλική τηλεόραση. Λοιπόν, 17 ε, Οκτωβρίου συναντηθήκαμε, 22 Οκτωβρίου τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών θεωρούνται δεκτά. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο 4 τώρα, το οποίο αφορά την έκβαση της συνδιαλλαγής στον προϋπολογισμό ε, του 13. Θα σας παρουσιάσω σύντομα την κατάσταση και μετά ε, θα ε, το παρουσιάσει το θέμα η εισηγήτρια Γένσεν. Η κυρία Χόλμαγερ ζητά συγγνώμη αλλά δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Πολλοί από εμάς, πολλοί από εσάς, Όλοι σχεδόν, εκτός από τον σκιώδη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πολύ κακό μαθητή, ο οποίος δεν ξενύχτησε μαζί μας, αλλά πάντως όλοι ήσασταν σχεδόν εκεί, στην τελευταία συνδιαλλαγή. Φυσικά το κοινό δεν ήταν ε, παρόν, απλά εκπροσωπήθηκε θα έλεγα και από τα άλλα όργανα. Ε, συμπερασματικά τώρα ε, κράτησε πάρα πολύ η συνδιαλλαγή, πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε κατ' εμέ. Και νομίζω ότι κάποια συμπεράσματα θα πρέπει να βγάλουμε από αυτό τώρα πλέον με ησυχία, με ψυχραιμία και να κάνουμε κάποιες συστάσεις και στους διαδόχους μας και στα άλλα θεσμικά όργανα γιατί ε, το να χρειαστεί κανείς 17 ώρες διαπραγματεύσεων άνευ διακοπής από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το πρωί έτσι ώστε να ανακαλύψουμε ότι η μέση οδός από το 0 στο 1 δις είναι 500 εκατομμύρια, αυτό είναι πραγματικά 16 ώρες και 30 λεπτά περισσότερο από όσο πρέπει. Οι, ε, αυτοί οι οποίοι θα έλεγα αγαπούν, ε, είναι ε, πραγματικά φίλοι των διαπραγματεύσεων, την καταβρήκαν σε εισαγωγικά, αλλά εγώ κουράστηκα. Και σας το λέω ότι βαρέθηκα λιγάκι και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν η τελευταία στην οποία πήρα μέρος σαν πρόεδρος, σαν εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου. Το τελικό αποτέλεσμα πάντως νομίζω και έρχομαι στην ουσία μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό απλά από το Κοινοβούλιο και γι' αυτό έγινε αποδεκτό από την αντιπροσωπεία την κοινοβουλευτική. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι συνθήκες, θυμίζω ότι η αντιπροσωπεία μας δεν ήταν μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ήταν μια αντιπροσωπεία η οποία συνετέθη από την διάσκεψη των Προέδρων, συνεστήθη, μάλλον από τη διάσκεψη των Προέδρων, για προφανείς λόγους οι περισσότεροι, τα περισσότερα μέλη ήταν μέλη της Επιτροπής μας. Και ε, υπεύθυνο για την αντιπροσωπεία αυτή ήταν κάποιος τον οποίο όρισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και θεωρητικά ο ίδιος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν ίσχυσε πέρυσι, ίσχυσε φέτος ο υπεύθυνος της αντιπροσωπείας, ο αρχηγός της αντιπροσωπείας υπογράφει επίσημα, διαχειρός, εξ του Κοινοβουλίου, όπως επίσης και ο εκπρόσωπος Υπουργός του Συμβουλίου Υπουργών. Και στη συνέχεια, το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης και συνδιαλλαγής υποβάλλεται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου είναι μια διαδικασία εντελώς διαφορετική και αποκλίνουσα από την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα για τον προϋπολογισμό του 2014. Η Επιτροπή μας δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει πλέον. Θα υπάρξει βέβαια μια ψηφοφορία. Η ψηφοφορία αυτή θα γίνει όμως στην Ολομέλεια και για το αποτέλεσμα της ε, ε συνδιαλλαγής και το αποτέλεσμα αυτό σύμφωνα με τα λεγόμενα της συνθήκης θα γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτός στην περίπτωση καταψηφιστεί η πρόταση από την πλειοψηφία των μελών που αποτελούν το Κοινοβούλιο. Εκτός δηλαδή αν υπάρξει μια ειδική αρνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Θυμίζω ότι σήμερα δεν θα ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του 2014. Θα ψηφίσουμε τον 9 διορθωτικό θα ψηφίσουμε επίσης ε, την χρήση του ε, οργάνου ευελιξίας ε, στην κατηγορία 2 και για την κατηγορία 1β για τη βοήθεια προς την Κύπρο που περιλαμβάνεται και στον προϋπολογισμό του 14. Η κατηγορία 2 ήταν ο διορθωτικός 7 και φυσικά θα γίνουν παρουσιάσεις και σχόλια για το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό το οποίο έλεγα. Προσωπικά θεωρώ ότι καταφέραμε να συνδυάσουμε δύο αντιφατικές μεταξύ τους απαιτήσει. Απαιτήσει όμως πολιτικής φύσεως και αυτό που λέω είναι θα έλεγα μια πολιτική αξιολόγηση. Κάθε μέλος και κάθε ομάδα φυσικά μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά νομίζω ότι μας επευλήθη η διαδικασία αυτή στο παρόν, στην παρούσα συγκυρία πολιτική και οικονομική. Λιτότητα δημοσιονομική καταρχάς. Λιτότητα σημαίνει καταρχάς νομική λιτότητα ένας ισορροπημένος προϋπολογισμός ο οποίος θα πρέπει να εκτελεστεί με ισορροπημένο τρόπο. Ο προϋπολογισμός του 13 αυτό ακριβώς θα κάνει. Και ο κίνδυνος τον οποίο διατρέξαμε το 2012 γιατί αν θυμάστε πατήσαμε λίγο την κίτρινη γραμμή για τον προϋπολογισμό του 14 με την θα έλεγα εφάνταστη σύλληψη έννοια των suspended payments, ε, των εναναβολή πληρωμών. Είχε τεθεί το θέμα, εάν πράγματι μπορούμε να αυξήσουμε τις πιστώσεις πληρωμών σε επίπεδο των ιδιαιτέρως υψηλών αναγκών του τελευταίου έτους και του τελευταίου έτους του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε αυτός ο κίνδυνος τελικά, λόγω ακριβώς της αυστηρής στάσης που κράτησε το Κοινοβούλιο, το οποίο την τελευταία στιγμή κατάφερε να πιέσει το Συμβούλιο και να αποκτήσει δύο δηλώσεις από πλευρά του Συμβουλίου. Πρώτον για την ανάγκη διαθεσιμότητας για αύξηση των πιστώσεων πληρωμών μέσω διορθωτικών προϋπολογισμών εφόσον πράγματι δημιουργηθούν ανάγκες για κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια υπέβαλε ε, την θετική ψήφο του για το πολιετές πλαίσιο στην σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για την αύξηση ε, κατά μέγιστον του ανωτά του ορίου για τις δαπάνες ε, ε, του 2013, το λεγόμενο Big Bang 11 δις 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα διέλθω τα διάφορα επεισόδια, το ότι χρειάστηκαν δύο φέτες ε, να κοπεί το πακέτο δηλαδή. Στην επιμονή μας για να πετύχουμε τη δεύτερη φέτα, το δεύτερο τμήμα, για τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το Συμβούλιο Υπουργών για να δεχτεί τα 3 δις 900 εκατομμύρια. Όλα αυτά ρυθμίστηκαν πλέον και θα πρέπει εδώ ε, εν παρόδο να πούμε ότι ήταν θετικό το ότι όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Κοινοβούλιο πέτυχε κατά το 2013 μία αύξηση θα έλεγα κατά 11, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τις ανάγκες τις πραγματικές ήταν κάτι το πάρα πολύ ικανοποιητικό. Καλό θα ήταν να ήμασταν ακόμα περισσότερο ικανοποιημένοι γιατί πράγματι σεβαστήκαμε τις συνθήκες, τηρήσαμε τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά οι αποδείξεις και οι λογαριασμοί που κλείνουν στο τέλος του χρόνου είναι αρκετά υψηλές και θα επιβαρύνουν και τον επόμενο. Αλλά από πλευρά της ικανότητα του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να στριμώξει το Συμβούλιο σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών νομίζω ότι αυτό που πετύχαμε ήταν σημαντικό. Ο Τζοβάνι δεν είναι ανάμεσά μας ή ίσως δεν είναι ακόμα ανάμεσά μας ο Τζοβάνι Λαβία, αλλά σε σχέση με την εκτέλεση του 2013, το τελευταίο κομμάτι, και ιδιαίτερα με τα έκτακτα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά από την πολιτική μας συμφωνία για το πολιετές πλαίσιο και για τα 11 δις 200 εκατομμύρια που είναι οι πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη με πολλά θύματα στη Γερμανία, στην Τσεχία, στη Ρουμανία και τα λοιπά και στην Αυστρία. Καταφέραμε παρόλα αυτά να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική διατύπωση 250 εκατομμύρια. Ανεβρέθησαν από τα 500, 509 εκατομμύρια του συνολικού, ε, της συνολικής πληρωμής και όχι 200 εκατομμύρια που είχε ψηφίσει το Συμβούλιο. Κάτι λοιπόν που μας επιτρέπει να έχουμε 100 εκατομμύρια επιπλέον από αυτά τα οποία ήθελε το Συμβούλιο. Για να μπορέσουμε να υπογράψουμε νέες συμβάσεις έρευνας και να διασφαλίσουμε την συνέχεια της πολιτικής βοήθειας στην έρευνα ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013. Για το 2014 το Συμβούλιο είχε μειώσει κατά ένα δις την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει τροπολογίες για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου δις, το οποίο ανταποκρίνεται με το ανώτατο όριο ε, του 2013 στο ανώτατο όριο του 13. Επιπλέον λοιπόν 150 ε, εκατομμύρια που προστέθηκαν στα 350 συνολικά μισό δις δηλαδή καλύψαμε το μισό της διαφοράς που είχαμε αρχικά. Θα ήταν βέβαια προτιμότερο να πετύχουμε το ένα δις αλλά στην παρούσα συγκυρία το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε δεν πρέπει να το υποτιμούμε και θα πρέπει η γραμματεία να μπορέσει να μας πει πότε πότε ήταν στο παρελθόν σε θέση το Κοινοβούλιο, πότε στάθηκε ικανό να αυξήσει τις πιστώσεις πληρωμών κατά μισό δις. Τα τρία τελευταία χρόνια ενθυμίστε ότι εμείς πολιτικά υποχρεωθήκαμε να δεχθούμε απόλυτα σχεδόν τις πιστώσεις πληρωμών που υπέβαλε το Συμβούλιο ενώ αυτή τη φορά μπορέσαμε να το αυξήσουμε κατά μισό δις. Ταυτόχρονα λοιπόν, από τη μία σεβόμεθα την λιτότητα όπως είπα και σε νομικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο και σε διαχειριστικό επίπεδο. Γιατί εάν τελικά συγκρίνουμε τον προϋπολογισμό στον οποίο καταλήξαμε μετά από την συνδιαλλαγή με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013 βλέπουμε ότι είμαστε 9 δις πιο κάτω. 6 με 7% λιγότερα χρήματα δηλαδή. Και νομίζω ότι κανένα από τα κράτη-μέλη δεν ψήφισε έναν προϋπολογισμό του 2014 που να μειώθηκε κατά 6 ή 7%. Και κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί να μας δώσει σε εμάς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαθήματα δημοσιονομικής λιτότητας. Κάποιοι το λυπούνται αυτό. Αυτό το οποίο είπα είναι πράγματι μια πολιτική εκτίμηση, αλλά έτσι είναι νομίζω. Και παρά αυτή τη διαπίστωση πετύχαμε, οι συγητές μας πέτυχαν να διευρύνουν εν πολλής τους πόρους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις οικονομικές προτεραιότητες και κυρίως στις κοινωνικές προτεραιότητες που καθόρισε το Κοινοβούλιο στην ψηφοφορία των τροπολογιών του τον μήνα Οκτώβριο. Προτεραιότητες οικονομικές ενισχύοντας με front loading πρόπληρωμες τα μέσα που έχει στη διάθεσή του το πρόγραμμα Horizon 2020, το COSME για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Erasmus και τις κοινωνικές προτεραιότητες τις οποίες θέσαμε με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νεωτέρων. Χάρη σε αυτή τη συμφωνία θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε στο επίπεδο που προεβλέπεται ήδη από το 2014 και θα αυξήσουμε ταυτόχρονα και τα προγράμματα για τη βοήθεια των ασθενεστέρων. Προσθέτω εγώ ότι καταφέραμε και εδώ η Γένσεν θα σας το πει με πιο αναλυτικό τρόπο να αυξήσουμε τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα η αύξηση αυτή φαίνεται ανεπαρκής εν πολλής, αλλά δυστυχώς ε, λειτουργήσαμε με περιορισμούς των ε, αρχών ε, εποπτείας, των οικονομικών αρχών εποπτείας, όπως επίσης και της εξωτερικής υπηρεσίας Frontex. Λοιπόν αυτά είχα να σας πω, αυτό θα μας οδηγήσει σε λίγο στο να υιοθετήσουμε τον προϋπολογισμό, τον διορθωτικό υπαρίθμε νέα ο οποίος θα θέσει ένα τέλος ε, στην δημοσιονομική διαδικασία εκτέλεσης, ε, την εκτελεστική δημοσιονομική του 13. Αλλά δεν θα ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του 14. Δίνω το λόγο στην Αν Γένσεν. Well, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δώσατε μια πολύ ωραία περιγραφή της κατάστασης και του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η κατάσταση. Δευτέρα προς Τρίτη σε αυτές τις 16 ώρες των διαπραγματεύσεων όπου για να είμαι ειλικρινής, για να είμαστε ειλικρινείς, οι διαπραγματεύσεις εξήγονται μεταξύ των μελών του Συμβουλίου των ίδιων. Και μερικές φορές είχαμε την εντύπωση ότι δεν ήταν ε, το Συμβούλιο παρόν στο, κτίριο ή ότι δεν είχαν ε, αντιληφθεί ότι είμαστε και εμείς παρόντες. Για να σας δείξω πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα στο Συμβούλιο αυτές, εκείνη την ημέρα, εκείνες τις δύο μέρες. Για ένα και μόνο αριθμητικό ποσό κατά βάση αυτών των πληρωμών. Και δεδομένων των δύσκολων συνθήκων στο Συμβούλιο, νομίζω μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα που πετύχαμε. Και τι νομίζω ανησυχούμε όλοι για την κατάσταση στις πληρωμές από εδώ και μπρος, δεδομένων των περιορισμών που υπάρχουν και είναι δεδομένοι και που μπορεί το 2014 να αντιληφθούμε ότι τα προβλεφέντα ποσά μπορεί να μην είναι επαρκή και γι' αυτό και για άλλη μια φορά ζητούμε δήλωση και δέσμευση από το Συμβούλιο πως όπως και εμείς άλλωστε δεσμευόμεθα θα προσφέρει στην Επιτροπή όταν χρειαστεί τα μέσα που χρειάζονται για να ικανοποιήσει τις απαιτήσει που θα έχουν οι πιστωτές εναντίτες για να εκπληρώσει υποχρεώσει Έχουμε λοιπόν σε σχέση με την ανάγνωση του Συμβουλίου 27 εκατομμύρια περισσότερα στην κατηγορία 1α, κυρίως για τα κοινωνικά προγράμματα και το ψηφιακό θεματολόγιο. Επίσης, στην ε, κατηγορία Α για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενισχύει, όπως είχαμε πει για το δημοσιονομικό πλαίσιο, ενισχύονται τα προγράμματα για την έρευνα, το Εράσμους, το κόσμο, το πρόγραμμα για την ε, καινοτομία. Στην κατηγορία 1Β έχουμε το Flex για το Κύπρο, και τα επιπλέον ε, κονδύλια για τις ε, μακροοικονομικές περιφερειακές στρατηγικές για τη Βαλτική και τις ε, νέες περιοχές που ανήκουν στο ζώνη του Δούναβη και προπαρασκευαστικές δράσεις. Στην δεύτερη κατηγορία, παροχή οπορικών στα σχολεία, ενισχύεται αυτό. Η Επιτροπή μας λέει ότι δεν θα υλοποιηθεί. Θα δούμε με τα ποσά που έχουμε ξεκινήσει, πώς, που έχουμε εξασφαλίσει, πώς θα προχωρήσει αυτό. Και στην κατηγορία 3. Στην κατηγορία 2 έχουμε το επίπεδο του ενός, έχουμε ένα ποσό ενός εκατομμυρίου για τη συμμετοχή στην Παγκόσμια Εκθέση στο Μιλάνο. Στην κατηγορία 3 έχουμε εξασφαλίσει τις, τις τα ποσά που θέλουμε για την ενημέρωση και πάλι ξεπερνούμε το ποσό που είχε προτείνει η Επιτροπή αρχικά. Όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάποιες άλλες ε, θέσεις στην κατηγορία 1α, ε, για τις οποίες όμως η Επιτροπή μας διαβεβαιώνει ότι μπορεί να τις ε, υλοποιήσει. Κατηγορία 4. Εξωτερικές σχέσεις, το μέσο ευελιξίας το προτείναμε εμείς, είχαμε ξεπεράσει το ανώτατο επίπεδο κατά 50 εκατομμύρια και γνωρίζαμε βεβαίως ότι αυτή η επιλογή θα ήταν δύσκολο να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο. Καταλήξαμε λοιπόν με ένα ποσό που είναι ακριβώς κάτω από το ανώτατο όριο, χωρίς όμως κανένα περιθώριο για την κατηγορία 4. Μόλις 400 εκατομμύρια έχουμε δηλαδή και το ποσό που είχε οριστεί για την Παλαιστίνη ε, που ήταν υψηλότερο από την πρόταση για το Συμβούλιο, του Συμβουλίου, α όχι, της Επιτροπής Αυτονομιλήτρια και έχουμε και 15 εκατομμύρια ευρώ πάνω από την πρόταση της Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Σε όλες τις υπόλοιπες ε, πιστώσεις που είναι προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο, και ε, ήταν προσεκτικά διατυπωμένη η συμβαστική πρόταση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Έχουμε ε, ποσά αναλογικά προς τη δική μας πρόταση. Χρειάστηκε λίγο να ε, την μειώσουμε για να είμαστε εντός των ορίων και να μείνουν ικανοποιημένες όλες οι πολιτικές ομάδες. Καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό, ο οποίος εξακολουθεί λοιπόν να ισχύει. Στον τίτλο 5 ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση. Ε, συζητήσαμε την υπόθεση του δικαστηρίου για το ζήτημα των μισθών και την ε, μισολογική ε, προσαρμογή. Θα δούμε τι θα βγει από αυτό. Θα είναι αρκετά μεγάλο το ποσό ενδεχομένως. Σε περίπτωση που χάσει το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσημειώσει κονδύλια προς την κατεύθυνση αυτή και προς το σκοπό αυτό και θεωρούμε ότι μπορούμε να το βάλουμε στο αποθεματικό αναμενώντας ε, την ε, απόφαση του δικαστηρίου. Έχουμε την κατάσταση όμως τώρα ότι δεν είναι στον κονδύλι, στη γραμμή του προϋπολογισμού εγγεγραμμένη αυτή η δαπάνη και θα χρειαστεί διορθωτικός ε, προϋπολογισμός εφόσον και όταν χάσει το Συμβούλιο στο δικαστήριο. Διότι μέχρι τώρα τι έχουμε δει ως ενδείξεις ότι μπορεί και να χάσει, είναι πιθανό να χάσει το Συμβούλιο αυτή την υπόθεση στο δικαστήριο πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Εκεί η συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο παραμένει ενισχύει, δηλαδή έχει αποφασιστεί. Για τους δορυφορικούς οργανισμούς agencies έχουμε έξτρα χρηματοδότηση ε, για το Frontex και το ASO. Ε, και την Ευρωπόλ για την καταπολέμηση ε, του εγκλήματος, γιατί έχουν νέες αρμοδιότητες για το ηλεκτρονικό έγκλημα τώρα στην Ευρωπόλ και χρειάζονται επιγόντως τα χρήματα αυτά. Και επίσης έχουμε και μια δήλωση που λέγει ότι θα πρέπει να συσταθεί ομάδα εργασίας ε, μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που να ορίζει πώς θα ανταποκριθούμε στις ε, ανακοινωθήσεις περικοπές κατά 5% τα έτη 2013 έως 2017 ως προς το προσωπικό. Γιατί έχουν μειωθεί ε, οι ώρες εργασίας και θα πρέπει να συνεχθούν τα θεσμικά όργανα πώς θα πετύχουν αυτό το στόχο και πώς η στελέχωση κάθε οργανισμού θα διαμορφωθεί στο μέλλον, διότι εμείς στο Κοινοβούλιο δεν συμφωνούμε με τα όσα πρότεινε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όσα έχει επιλέξει ως ε, λύση ότι οι οργανισμοί που αυξάνονται ε, να παίρνουν αυτόματα προσωπικό και να στελεχώνονται από προσωπικό άλλων οργανισμών που μειώνονται. Είναι και πολιτικές οι αποφάσεις για να δούμε κατά πόσο η στελέχωση είναι σωστή και οικονομική πόρη. Ε, για να ανταποκρίνονται στο καθήκον που τους έχουμε αναθέσει οι διάφοροι οργανισμοί. Δεν μας πειράζει μας να γίνουν περικοπές, αλλά όχι αυτόματα και οριζόντια στους οργανισμούς. Εάν θέλουμε περικοπές, να δούμε τις ιδιαιτερότητες και να δούμε κατά πόσο συγχωνεύονται, ενδεχομένω οργανισμοί κλείνουν, να είναι πιο αποτελεσματική λειτουργία, αλλά όχι με οριζόντια μέτρα και να μην προσπαθούμε να τους στραγγαλίσουμε σταδιακά και ε, αργά αλλά σταθερά για να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά ήταν τα βασικά που ήθελα να σας πω και γενικά πιστεύω ότι καταφέραμε τις περισσότερες προτεραιότητες μας να τις ε, επιβάλλουμε. Ξέρετε, είναι συμβιβασμός αυτό. Και δεν είμαστε και σε πάρα πολύ ισχυρή θέση, διότι Ε, δεν ήταν λύση η άλλη λύση με τα 12 τιμόρια, ε, το να μην υπάρχει καθόλου προπολογισμό και θεωρήσαμε ότι ήταν και δική μα ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ε, προπολογισμό. Μέσα σε αυτό το πολύ στενό χρονικό πλαίσιο που είχαμε στη διάθεσή μας και στην πολύ δεινή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Θα ήθελα με ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την τους, επικοδομητική συνεργασία. Νομίζω ότι είμαστε μια πολύ συνεκτική ομάδα. Παρόλο που ορισμένοι δεν ε, συμφώνησαν με τη γραμμή της πλειοψηφίας, πάντως ε, είχαμε μια σοβαρή και καλή ανταλλαγή απόψεων. Και είχα επίσης την αίσθηση ότι η Λιθουανική Προεδρία πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε για να βεβαιωθεί ότι θα γίνει η συζήτηση με τρόπο ειλικρινή και ανοιχτό. Ήξεραν και εκείνοι ποιες είναι οι δικές μας κόκκινες γραμμές και εμείς τις δικές τους. Και θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν ένα ειλικρινής και τίμης διαμεσολαβητής που είναι σημαντικό και αυτό για να υπάρξει ένα ειρηνικό αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το να χρειαστεί να περιμένουμε 12 ώρες για να έρθει η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου ήταν πάρα πολύ και συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι κάποιος θα πρέπει να προβληματιστεί για σε αυτό το θεσμικό όργανο. Αν είναι πραγματικά ένας τρόπος αξιοπρεπής να εργαζόμαστε και να χειριζόμαστε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Περάσαμε μια βραδιά ολόκληρη μαζί αυτό έχει τις χαρές του και τις χάρες του. Αλλά βέβαια ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη για τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ Άννα. Ο Τζοβάνι δεν είναι εδώ. Αλλά ο Σαλβαδόρ Γκαρίγκα μας έχει στήσει το λόγο. Πολύ σύντομα. Διότι συμμερίζομαι όλες τις εξηγήσει που έδωσε η Άν και τη συγχαίρω προσωπικά την ίδια αλλά και τη Μόνικα Χολμάιερ οι συγκίτριες του προπολογισμού και του γενικού αλλά και των ε, λοιπόν ε, οργάνων για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα, διαπραγματεύτηκαν και υπερασπίστηκαν τις θέσεις του. Πράγμα που κατέστησε ενδιαφέρουσα τη συνεδρίαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πραγματικά εξέθεσαν ποια είναι τα όρια του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης ε, να ε, συγχαρώ όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας που αντέξατε τόσες ώρες και να τονίσω ότι ένα από τα κληροδοτήματα που θα πρέπει να αφήσουμε στους συναδέλφους που θα έρθουν με το καλό του χρόνου τέτοιο καιρό να αντιμετωπίσουν τη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό, ότι αυτός ε, ο τύπος συνδιαλλαγής είναι τελείως παράλογος. Δεν μπορεί να κάθεσαι τώρα 18 ώρες στο κτίριο του Συμβουλίου να περιμένεις μια απλή συνεδρίαση επειδή χρειάζεται ε, το Συμβούλιο όλες τις διαφορετικές ε, συνεδριάσεις να τις κάνει διμερείς. Το Κοινοβούλιο είναι ευέλικτο και μπορεί σε μια συνεδρία μισή ώρα να λύσει το θέμα και να αντιδράσει στι αλλαγέ των διαφόρων θέσεων. Αυτό το σύστημα μου φαίνεται τελείω παράλογο και νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε όχι εμείς και το Συμβούλιο για ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο να καταλήγουμε σε αυτή τη συνδιαλλαγή. Ένα ίσονο σημασία θέμα, μια λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής νομίζω ήταν το καλύτερο δυνατό σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για όλα τα κράτη-μέλη. Το 2013 είναι ε, έτος ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης σε όλα τα κράτη-μέλη, οπότε οι ταμιακές ε, δυνατότητες είναι παντού σφιχτές σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είχε σημασία όλη η διαδικασία του 2013 που είναι και πάλι καρπός της ε, προηγούμενης διαδικασίας του 2012 που ναυάγησε. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, ακριβώς επειδή ναυάγησε η συνδιαλλαγή δεν θα είχε κινητοποιηθεί αυτή η διαδικασία και θέλω να ευχαριστώ σε όλους ιδιαίτερο τον πρόεδρο Λαμασούρ για την πρωτοβουλία του να τεθεί ακριβώς σε ένα πραγματικό σύστημα ε, ανείχνευση στο πώς ακριβώς έχουν οι πληρωμές και τι χρειάζεται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τα επόμενα έτη. Από την άλλη πιστεύω ότι συνεισφέραμε κι εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι στη θέση που της αξίζει. Δηλαδή να παρέχει τους πραγματικούς αξιόπιστους και σαφείς αριθμούς και τα στοιχεία για το ποιες είναι οι ανάγκες της πιστώσης πληρωμών. Και έτσι φέτος αποφύγαμε το περσινό πρόβλημα όπου το Συμβούλιο διαρκώς αμφισβητούσε και απέριπτε τα αριθμητικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φέτος αυξήσαμε βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να αυξηθεί η αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων και όπως είπαν και οι συνάδελφοι για πρώτη φορά το Συμβούλιο αναγκάστηκε να δεχτεί ότι χρειάζεται να ε, τροποποιήσει και να αναθεωρήσει προς τα πάνω τους υπολογισμούς. Γιατί, Γιατί κατάλαβε ότι είναι αξιόπιστα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ανέβηκε και στην εκτίμηση ε, και στην αξιοπιστία και στο κύρος. Αυτά. Νομίζω ότι τελειώσαμε τη θητεία αυτή βάζοντας τα θεμέλια για το μέλλον και προτείνοντας ένα σύστημα επαλήθευσης των πραγματικών στοιχείων ε, πληρωμών που χρειάζονται θεσμικά όργανα για να λειτουργούν και αυτό είναι καλό και για τους φορολογούμενους αλλά και για τη δημοκρατική διαφάνεια των θεσμικών οργάνων. Και συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Euh, euh, Ευχαριστώ ο βγήκε για να μην ακούσει ο Λαδόρ και τώρα ξαναγυρνάει από ό,τι φαίνεται για να πει τα δικά του. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι την ουσία και τα πιο σημαντικά του Σαλβαδόρ τα έχω υπόψη μου. Θα ήθελα απλώ να πω ότι βεβαίω και υποστηρίξαμε την ε, συμφωνία και τη συνδιαλλαγή και το κοινοβούλιο είχε ε, σημαντική ρόλο να δραματίσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να πούμε ότι εφέτος οι εκρεμείς πληρωμές θα περάσουν στο 2014, όπως άλλωστε και τα επίπεδα των πληρωμών που έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο είχε ε, μείνει σε ποσά πολύ χαμηλότερα από αυτά που είχε προτείνει η Επιτροπή. Και έτσι πιστεύω ότι του χρόνου με πολύ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να υπαγρυπνούμε ώστε να μην ε, ε, χαθούν οι προτάσεις της Επιτροπής Κρατών Μελών και να μην καθυστερήσουμε πολύ την ε, λειτουργία των προγραμμάτων λόγω ελλείψεως σπόρων. Ευχαριστώ πολύ Βάιλο, έχεις πολύ το δίκιο. Η ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ζήτησα το λόγο για να συγχαρώ την εισηγήτριά μας για όλο της το έργο, όλο αυτό το χρόνο. Ήταν αρκετά περίπλοκη όλη αυτή η υπόθεση. Γιατί μπορεί να έχει αρχίσει να εργάζεται στον προπολογισμό από τον Ιανουάριο. Υπήρξαν καθυστερήσεις με συμφωνίες για το πολιτισμικό δημοσιονομικό πλαίσιο κτλ. Και τελικά ήταν μια κούρσα ε, όλη αυτή η υπόθεση και μάλιστα ασαφή ε, και αβέβαιη έκβαση. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν αρκετά απλή, διότι είχαμε κάποια περιθώρια που μας εμπόδιζαν να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι στην ανάγνωση του προπολογισμού, αλλά τελικά νομίζω ότι η συμφωνία μπορεί κάλλιστα να γίνει ε, αποδεκτή. Όπως είπε όμως και ο Βάιλο, το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι δεν έχει λυθεί το θέμα των πληρωμών. Για πρώτη φορά είναι γεγονός. Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να αυξήσουμε τις πληρωμές 500 εκατομμύρια ευρώ και καλώς να ορίσουν. Αλλά είμαστε γύρω στα 20 δις ε, τιμολογίων που δεν έχουν εξοφληθεί. Και όταν ε, φτάσει η ώρα ε, να αρχίσουμε να πληρώνουμε και να φτάνουμε σε αυτή την οροφή το ανώτατο όριο πληρωμών, θα πρέπει το, θέμα να το δει το Συμβούλιο. Και δεν ξέρω τι τους κληροδοτούμε ε, στους συναδέλφους του επόμενου Κοινοβουλίου ακριβώς. Ελπίζω μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή να το σκεφτεί και το Συμβούλιο και να κοιτάξει με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα όταν το βρει μπροστά του. Γιατί αυτή τη στιγμή ανησυχώ και από τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου, το οποίο αποπειράθηκε να διευκρινίσει τη δική του ανάγνωση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ειδικά μέσα και προσπάθησε να πει ότι μιλάμε για συμβιβασμούς και για άλλη μια φορά απέφυγε το ποτήρι των πληρωμών. Και κάτι άλλο ε, που μας βρίσκει όλους συμφωνούς είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συνδιαλλαγή. Δεν μπορεί να διαρκεί 17-18 ώρες. Είναι απαράδεκτο. Και για το Κοινοβούλιο η πραγματική διάρκεια των διαπραγματεύσεων πόσο ήταν, δύο ώρες, ούτε καν. Εμεί τι κάναμε, περιμέναμε να δεήσει, να συμφωνήσει το Συμβούλιο με κάποια πρόταση. Και μετά από ένα δωδεκάωρο ή δεκάωρο ήρθε η πρώτη πρόταση που ήταν τελείω μακριά και από την πραγματικότητα και από οποιαδήποτε αποδεκτή και παραδεκτή θέση για το Κοινοβούλιο. Κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο τρόπο λειτουργία του Συμβουλίου, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν 28 χώρε με 28 πραγματικότητε και 28 διαφορετικού στόχου. Ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε ως 18 ώρες να συμβεί κάτι τέτοιο. Μήπως αρχίσει κάποια στιγμή η συζήτηση με το Συμβούλιο. Γιατί και για εκείνους νομίζω θα ήταν ε, εύστοχο και σκόπιμο να γίνει μια τέτοια συζήτηση για το μέλλον. Πώς θα πάμε στις συνδιαλλαγές. Έχουμε ευτυχώ εξέλιξη στην τεχνολογία, νέα εργαλεία. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε στην ίδια αίθουσα η μεν δε. Και η πραγματική συνδιαλλαγή δεν μπορεί να γίνει την τελευταία μέρα από τις 21 μέρες που έχουμε για τη συνδιαλλαγή. Υπάρχουν πολλές μέρες που μπορούμε να επιμερίσουμε την εργασία, να συμπλησιάζει τις θέσεις στο Συμβούλιο και όταν φτάνουμε στο παραπέντε της συμφωνίας να συναντιόμαστε όλοι και να οριστικοποιούμε τη συζήτηση. Δεν μπορούμε 18 ώρες να διαπραγματευόμαστε γιατί έχουμε και τα βιολογικά μας όρια. Και δεν είναι πραγματικές αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αυτό και μόνο θα πω. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριος Μίλτος. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτα ικανοποιημένος βεβαίως. Το έχω πει και άλλες φορές, έτσι συμβαίνει και με την παρούσα συμφωνία, αλλά υπάρχουν πολύ διαφορετικέ απόψει και συμφωνώ με όλου εκείνου που λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε από τι παρούσε συνθήκε να εξασφαλίσουμε. Φυσικά πρέπει να υπογραμμίσουμε επανειλημμένω ότι αυτό ο προπολογισμό είναι κατά 6,5% ε, μικρότερος, χαμηλότερο από αυτόν του προηγούμενου έτου. και θα ήθελα να μου πει κανεί αν υπήρξε ποτέ Εθνικό Κοινοβούλιο το οποίο να έχει επιτύχει αντίστοιχη μείωση σε εθνικό προπολογισμό. Και αυτό και αυτό εν βεβαίως και των ευρωεκλογών και της ιδέας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ξέρει να δείχνει οικονομία στη διαχείριση των κονδυλίων. Νομίζω ότι υπό το φως της λιτότητας μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε όπως και άλλοι. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Αν που παρακολούθησε με τον λεπτό και διακριτικό της τόπο πάντα τις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν την είδα ποτέ ούτε εκνευρισμένη, ούτε θυμωμένη, ούτε οργισμένη. Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ε, γιατί το να, περιμένει κανείς το Συμβούλιο για ατελείωτες ώρες ε, χωρίς ε, καμιά άλλη επιλογή μπορεί να δοκιμάσει και τα πιο γερά νεύρα. Όπως υπόθηκε πάντως, το σημαντικό στοιχείο είναι πληρωμές. Το Συμβούλιο πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν αρκεί να αναλαμβάνει δεσμεύσεις υποχρεώσεων, αλλά λαμβάνει υποχρεώσει, αλλά και να τις εκπληρώνει, να τις καταβάλει. Αυτό. Πρέπει να το τονίσουμε. Πάντα στο τέλος της εκτέλεσης ενός προπολογισμού μένουν διαφωνίες και διαφορές για το τι ε, πρέπει να πληρωθεί, τι πρέπει να εξοφληθεί μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής αλλά και Κοινοβουλίου επίσης. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι είναι ουσιώδες για να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα και λειτουργία του προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Άλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω ορισμένε παρατηρήσει. Λένε ορισμένοι αλήθεια, ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο δυνατό εάν αυτό είναι το καλύτερο δυνατό. Δεν ήμασταν και τόσο θραλέοι. Ούτε και τα καταφέραμε τόσο καλά. Δεν πετύχαμε τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή. Η πολιτική μου ομάδα δεν συμμερίζεται την αισιόδοξη ή λιγότερο απεσιόδοξη ανάγνωση της καταστάσεως στην οποία έχουμε από τις άλλες ομάδες. Νομίζω ότι υπολοιπόμεθα σημαντικά των προσδοκιών και ελπίδων του Ευρωπαίου πολίτη και υπολοιπόμεθα πολύ και των προοπτικών που είχαμε εμείς ως Κοινοβούλιο ορίσει για τον Ευρωπαίο πολίτη, διότι έχει τις προσδοκίες του πολίτης, οι οποίες προσδοκίες εκφράζονται με δεσμεύσεις ε, διαδοχικές, ότι θα στηρίξουμε τους νέους, ότι θα τους προσφέρουμε προγράμματα απασχόλησης, ότι θα τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας, ε, ότι η έρευνα και η καινοτομία θα αποτελέσουν ευκαιρίες για εξέβρεση εργασίας και τελικά το αποτέλεσμα, στη, συγκρινόμενο με τις προσδοκίες που είχαν καταργηθεί στον ε, Ευρωπαίο πολίτη, είναι πολύ ισχνό. Με προϋπολογισμό με βάση τους δικού σα κατά 6% χαμηλότερο, αλλά μπορώ να σας πω ότι αν είχαμε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού, ε, ότι ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού θα μα οδηγούσε σε αποτέλεσμα κατά 9% χαμηλότερο από τον προηγούμενο προπολογισμό. Είναι προφανώ ανεπαρκέ το αποτέλεσμα λοιπόν και εν γέννη λέγεται ότι εάν ξαπλώνει κανεί και προσπαθεί να σκεπαστεί με μια κουβέρτα που του πέφτει πολύ, με ένα πάπλωμα που του πέφτει πολύ κοντό, ή τα πόδια του θα κρυώσουν ή η η του. Όταν λοιπόν έχουμε ένα προπολογισμό τόσο ισχνό, προφανώς κάποιες από τις ε, δράσεις δεν θα υλοποιηθούν αφού δεν αρκούν τα χρήματα. Κατά τα άλλα, ναι, βλέπουμε μια μικρή αύξηση στον ε, τομέα της έρευνας, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το Εράσμους, όπως βλέπει τα πράγματα του Συμβούλου τουλάχιστον, αλλά πρόκειται για αυξήσεις οι ε, και μάλιστα για αυξήσεις οι οποίες προέρχονται από την ε, μεταφορά κονδυλίων προς τον προϋπολογισμό, πράγμα όμως το οποίο δεν ε, εξασφαλίζεται με τον ίδιο τρόπο στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει πρόγραμμα για την ενίσχυση των πιο στερημένων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Κοινωνικού Ταμείου και ο αγώνας, η καταπολέμηση της ενεργείας των νέων που θα καταπολεμηθεί από τα, ε, θα χρηματοδοτηθεί από τα ε, διάφορα κονδύλια που αναπτύσσονται κατά περιφέρεια. Για την, ανα... για την ανθρωπιστική βοήθεια έχουμε μπορέσει εμείς ως Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουμε αύξηση των ποσών σε σχέση με αυτά που πρότεινα το Σύμβουλο και η Επιτροπή και χαιρόμαστε ιδιαίτερως, αλλά δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των προσφύγων όπως θα έπρεπε και το πρόσφατο ε, τραγικό ατύχημα στη Λαμπεντούζα συγκλώνησε τους πάντες, πολίτες όσο και βουλευτές. Ωστόσο, όταν, εάν αναζητήσουμε το πώς εκφράζεται αυτή η ανησυχία ε, σε όρους δημοσιονομικούς, μόνο μια πολύ μικρή αύξηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για το άσυλο βλέπουμε να δίδεται και μια αύξηση ε, ισχνότατη μόλις τα 2 εκατομμύρια για την ε, Frontex. Για την ομάδα μου λοιπόν το πρόβλημα των ε, προσφύγων, των τραγωδιών όπως αυτό της Λαμπετούζα δεν μπορεί να ρυθμιστεί από τη Frontex και τις αστυνομικές αρχές. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να ρυθμιστούν τα προβλήματα αυτά. το Ταμείο για το Άσυλο είναι υποχρηματοδοτούμενο. Δεν, δεν αρκούν τα κονδύλια που έχουν προβληθεί. Για να ολοκληρώνω, ο υπολογισμό αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα στο πολυεθνικό συνομικό πλαίσιο, αντικατοπτρίζει λιτότητα και περικοπέ. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει την ανατροπή της λιτότητας, ούτε βέβαια και στη λύση, στη διέξοδο από την ανεργία. Για τα λοιπά, και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, η διαδικασία που πρέπει να αποδεχθεί κανείς έχει ή μη τι άλλο στοικό χαρακτήρα ή αλλιώς θα έλεγα και μαζοχιστικό γιατί πρέπει να περιμένει κανείς ώρες ατελείωτες και εύχομαι καλό κουράγιο σε όποιον αναλάβει τα ενία αργότερα. Ένας Άγγλος χιουμορίστας είπε ότι ο αισιόδοξο είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Το ίδιο και ο απεσιόδοξος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το αποτέλεσμα για το προϋπολογισμό του 2014 ευτυχώς μετά ε, τη στάση του Συμβουλίου είναι λιγότερο κακό από όσο θα επιθυμούσε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά για τους πολίτες είναι χείριστο το αποτέλεσμα δυστυχώς και παραμένει. Και θα παρακαλούσα το Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση και θα είναι βούτυρο στο ψωμί μας ε, ε, υπέρ του ευρωσκεπτικισμού. Και πρέπει να σας πω ότι το κόμμα μου και εγώ θα καταψηφίσουμε αυτό τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την επεξήγησή σας. Λοιπόν, συνάδελφοι, αυτά είχαμε να πούμε για τον προϋπολογισμό των τον των υπαρίθμεν όπως επίσης και τον κανονικό προϋπολογισμό για το 2014. Τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα αναφερθούμε στην πρώτη ψηφοφορία την οποία θα κάνουμε, η οποία αφορά τον κανονισμό για το πολιετές πλαίσιο. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε συνάδελφοι τώρα, θα ψηφίσουμε πρώτα τον κανονισμό για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θα ήθελα ένα άλλο θέμα. Είχαμε πει εξ αρχής ότι δεν θα συμφωνούσαμε με τα πάντα, αν δεν είχαν συμφωνηθεί τα πάντα. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες για τους ιδίους πόρους υπάρχει η Επιτροπή η οποία το συζητά αλλά επίσημα ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Και νομίζω ότι η διαδικασία δεν είναι ικανοποιητική. Αν κατάλαβα καλά, χθε το απόγευμα έγινε μια διάσκεψη των Προέδρων και αποφάσισαν ότι το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα θα τεθεί ε, στην ημερήσια διάταξη της επόμενης εβδομάδας με αστερίσκο. Αν δεν έχουμε δηλαδή ε, πληροφορίες για μια κάποια επιστολή από την Επιτροπή κτλ. δεν θα προχωρήσουμε. Σήμερα το πρωί από κάποια, ε, με κάποιο μυστήριο τρόπο αφαιρέθηκε ο αστερίσκος και το θέμα αυτόματα μένει στην στην ψηφοφορία, για ψηφοφορία στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Η διαδικασία λοιπόν δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Εγώ θα ήθελα να παραμείνει ο αστερίσκος στην α, ημερήσια διάταξη επίσημη προϋπόθεση για να πάρουμε μέρος στην ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ Γιάννα. Νομίζω και εγώ τα ίδια ήθελα να πω θα με προκαταλάβεις και εσύ και ο Ιβάιλο και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Γιάν λέει ο Ιβάιλο. Ο Αλφονσί, για το συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζω ότι οι μεγάλες ομάδες θα δεχθούν το νέο δημοσιονομικό και πράγματι όταν είμαστε υπεύθυνοι για μια παράδοση ουσιαστικά ανεφόρων θέλουμε να ξεμπερδεύουμε. Πάντως νομίζω ότι στο θέμα των ιδίων πόρων είναι πολύ σημαντικό και εξαρτάται από αυτό η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν ζητήσαμε εμείς με το ψήφισμά μας από την ομάδα, να δημιουργηθεί η ομάδα εργασίας, η Επιτροπή Εργασίας, στην ουσία θέσαμε εν κινδύνο, αν θέλετε, ένα τμήμα της αξιοπιστίας του Κοινοβουλίου. Ίσως να υπάρχει μια καθυστέρηση τυπικού χαρακτήρα, οπότε η Επιτροπή θα κάνει την πρότασή της την επόμενη εβδομάδα και τη Δευτέρα ε, θα ψηφίσουμε. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Θυμίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Είδαμε ότι φέτος μειώθηκαν ε, λόγω των λιγότερων εισπράξεων από τα τελωνία. Υπάρχουν συμφωνίες ε, για τη Λατινική Αμερική που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο τους πόρους αυτούς και δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε την επιτροπή, δεν έχουμε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, δεν έχουμε τον οδικό χάρτη. Θα ήταν πράγματι πολύ ελαφρύ από πλευρά μας να δεχθούμε μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να αναβάλουμε την πληροφορία. Και αν η ψηφοφορία δεν μπορέσει να γίνει τον Νοέμβριο, να γίνει το Δεκέμβριο, μέχρι ότου έχουμε όλες τις εγγυήσεις που απαιτείται. Κοιτάξτε, δεν θέλω να γίνει μια συζήτηση εκ νέου για το θέμα αυτό. Έχουμε μιλήσει για τα θέματα αυτά επί μακρόν. Ας μην λέμε ότι δεν έχουμε καμία εγγύηση για την ομάδα α, υψηλού επίπεδου. Το μοναδικό πολιτικό πρόβλημα για την ομάδα αυτή, πάνω στο οποίο ε, εργάζομαι σκληρά εδώ και έξι μήνες, Ε, πράγματι αν δεν υπήρχα εγώ δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτή η ομάδα και συγγνώμη που το λέω έτσι εγωιστικά. Αλλά το πρόβλημα το πολιτικό είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία για το πρόσωπο που θα προεδρεύσει αυτής της ομάδας. Γιατί, γιατί οι μεγάλοι αρχηγοί δεν το συζήτησαν. Ένας πρόεδρος ομάδας έκανε μία πρόταση, πρότεινε ένα όνομα, εγώ προσωπικά επίσης σε προσωπικό επίπεδο πρότεινα και κάποιες άλλες. Οι δικές σας ομάδες δεν έχουν κάνει προτάσεις και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στην τελική διατύπωση των μεθόδων εργασίας, τις σχέσεις με τα όργανα και το χρονοδιάγραμμα, εφόσον δεν έχουμε το όνομα του προσώπου που θα ηγηθεί, που θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο υψηλού επίπεδου, για να προεδρεύσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Αν βάλουμε έναν υψηλό βαθμό υπάλληλο, τότε θα έχουμε χαμηλό βαθμό υπαλλήλου σαν μέλη της ομάδας. Αν βάλουμε έναν τέος αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης, τότε η ομάδα αυτή θα είναι σε υπουργικό επίπεδο, πάρα πολύ απλά. Και αυτό το, αυτή η προσωπικότητα θα έχει πολλά να πει και σημαντικά για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί η ομάδα έχουμε φτάσει στο απότατο χρονικό όριο του τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών. Υιοθετώ λοιπόν την παρατήρηση του Γιάννα που υποστήριξε και ο Ιβάιλο. Εμείς οφείλουμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όταν πράγματι ε, αποφασίσουμε με την ψηφοφορία μας στην Ολομέλεια, στην Ολομέλεια τελικά για το πολιετές να έχουμε τις απαραίτητες εγγυήσεις. Ε, ευχαριστώ τη Λιθουανική Προεδρία η οποία είναι παρούσα, ας εξέφρασα την εκτίμησή μου για σας αλλά δεν ήσασταν παρούσα. Ε, είδαμε που βρίσκονται οι εργασίες στο Κορεπέρ, δεν είναι ικανοποιητικές και θα πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων να το επανεξετάσει. Όπως ακριβώς το είπε και ο Γιάν Μούλτερ θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αστερίσκος θα μπορέσει να υπάρξει και αναβολή. Πρέπει όμως τώρα να ψηφίσουμε εμεί σε επίπεδο Επιτροπής Προϋπολογισμών γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέραν αυτού το οποίο θα κάνουμε. Αν δεν ψηφίσουμε σήμερα δεν θα ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς την επόμενη εβδομάδα. Αν δεν ψηφίσουμε σε επίπεδο δηλαδή Επιτροπής οι προθεσμίες αυτό δείχνουν. Λοιπόν έχετε υπόψη σας έτσι έχουν τα πράγματα και είχαμε κι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο είχε οδηγήσει τους ίδιους άλλωστε να ζητήσουν αναβολή και το είχα δεχτεί γιατί ήταν απόλυτα θεμητό. Ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να ελέγξουμε από πλευρά μας. Το ελέγξαμε με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κείμενο λοιπόν του άρθρου 8 του κανονισμού MFF θα πρέπει να διορθωθεί για να είναι συμβατό με το άρθρο 21 του κανονισμού των Ταμείων Συνοχής Έχετε λοιπόν στο Κόμπου News το κείμενο έχει κυκλοφορήσει, σας το διαβάζω στα αγγλικά, λέγεται ότι στην περίπτωση ε, απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο, τα Ταμεία Συνοχής, το ΦΕΟΓΑ ή το Ταμείο, εν πάση περιπτώσει, Αλληλείας και Ναυτιλίας, ε, που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ταμείων αυτών με μια σωστή οικονομική διαχείριση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μεταφέρει τις πιστώσεις που δεν έχουν καταβληθεί στον επόμενο χρόνο, που δεν θα πρέπει να ε, είναι διαθέσιμα ε, σύμφωνα με τον κανόνα 1 συν 3. Το άρθρο λοιπόν 10 του κανονισμού τροποποιήθηκε με βάση τη νέα διατύπωση του άρθρου 8 και η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων συμφωνεί με το κείμενο αυτό και γι' αυτό και το εισάγαμε. Λοιπόν, αυτά θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για το MFF. Θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν τον δημοσιονομικό ε, πλαίσιο για τον κανονισμό δημοσιονομικού πλαισίου ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α, έχουμε και τροπολογίες, ζητώ συγγνώμη. Α, έχουν μοιραστεί τροπολογίες. Λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία πρώτα τις τροπολογίες. Τέσσερα της κυρίας Τρούπελ, εισηγητής κατά ποιοι είναι υπέρ. Τέσσερις, ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία α και β των εισηγητών από κοινού. Είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 5. Φερέιρα. Ε, έχουμε πολλούς Φερέιρα του κυρίου Φερέιρα. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. κατά απορρίπτεται η, πέντε τώρα η ένα της κυρίας Τρούπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 η συγητής είναι υπέρ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 3 των φιλελευθέρων. Ο είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τελική ψήφος ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έχετε όλοι πέρας της ψηφοφορίας 28 υπέρ, 5 κατά, 0 αποχές, δεκτή η πρόταση κανονισμού. Έχουμε τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία της επιβεβαίωσης του ένατου ε, διορθωτικού. Μία ψήφος, δεν έχετε κατάλογο εδώ να, για να ψηφίσετε γιατί υπάρχει μία και μόνη ψηφοφορία. έτσι ώστε να υπάρξει ταύτιση και με την πρόταση του Συμβουλίου μέσω της προφορικής τροπολογίας της σοσιαλιστικής ομάδας η οποία έχει διανεμηθεί και η οποία λέγει ότι το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι παραμένει στη θέση αρχής του ότι η χρηματοδότηση μέσων όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό πέρα των ορίων του πολιετούς πλαισίου και οι δηλώσεις μονομερής του Συμβουλίου ε, θα προσαρτηθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2014. Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι αυτό που ονομάζουμε στη γαλλική γλώσσα ανταπόδοση. Γιατί στις 4 ώρα το πρωί, τη στιγμή που υπογράψαμε την, ε, ε, την συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια μονομερής δήλωση του Συμβουλίου, η οποία λέει ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο όλα τα μέσα ευελιξίας τα οποία είναι προσαρτημένα στο MFF θα πρέπει να μείνουν κάτω από το όριο. Εμείς δεν μπορούμε να εμποδίσουμε βέβαια το Συμβούλιο να κάνει μονομερείς δηλώσεις ακόμα και αν είναι ανόητες. Και το Συμβούλιο δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να το κάνουμε ούτε εμείς το ίδιο. Για να συνεχίσουμε λοιπόν το παιχνίδι, λέμε ακριβώς μέσω της προφορικής μας τροπολογίας ότι η δήλωσή τους είναι ανόητη και ότι η δική μας ερμηνεία είναι η σωστή. Αυτό θα δώσει στους διαδόχους μας τροφή για συζήτηση. Για τον διορθωτικό αυτό προϋπολογισμό μέσω της προφορικής τροπολογίας ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας, 33 υπέρ, 2 κατά 0 αποχές δεκτό. Έχουμε μια τελευταία ψηφοφορία, ε, ομαδική θα έλεγα, είναι η έκθεση Ντεάννα για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για τη βοήθεια προς την Κύπρο. Όχι, δεν μπορεί να γίνει δια ανατάσεως ε, το Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Το σύστημά μας ε, είναι ε, γραμματιοκεντρικό. Η γραμματεία αποφασίζει. Εν πάση ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την Κύπρο. Παρακαλώ κινητοποιηθείτε. Πέρα στις ψηφοφορίες ψηφίσατε όλοι. 33 υπέρ, 2 κατά. 0 αποχές. Οι δύο τελευταίοι που ξύπνησαν και ψήφισαν καταψήφισαν. Λοιπόν δεν τελειώσαμε όλες τις ψηφοφορίες, αλλά τελειώσαμε τις ψηφοφορίες τις σχετικές με το πολιετές πλαίσιο και με τον προϋπολογισμό. Στην παρούσα φάση ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών λέει αρκετά. Ουφ. Απαλλάχτηκα. Να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και για το πολιετές πλαίσιο και για τον προϋπολογισμό και για τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς του 2013, έστω και τη απουσία τους. Την εισηγήτρια για τους εισηγητές μάλλον για το προϋπολογισμό του 14 και τη Χωμάγερ που δεν είναι εδώ και κυρίως την Άννα. Τεράστια δουλειά και μεγάλη επιτυχία αυτό για τη Γένσεν η οποία ολοκληρώνει την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς για το Κοινοβούλιο δεν σκοπεύει να ξανάρθει. Θα ήθελα παρακαλώ να χειροκροτήσουμε τη Γένσεν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Λιθουανική Προεδρία όλους ιδιαίτερως, τον Υπουργό και εκείνο αξίζει συγχαρητήρια. Τον Υπουργό, τον Πρεσβευτή, ε, εμάς τους ιδίους, τον Προεδρεύοντα της ομάδας του Συμβουλίου για τον Προπολογισμό, επισήμως είσαστε οι εχθροί μας. Φέρνουμε σε αντιπαράθεση δηλαδή τις θέσεις των θεσμικών οργάνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως απαιτεί να γίνεται αυτή η αντιπαράθεση και τη γεγονό ότι καταλήξαμε στη συμφωνία αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ότι έγινε καλή δουλειά και από τις δύο πλευρές και θα ήθελα να ευχαριστώ την Προεδρία της Λιθουανίας. Και μια και δεν έχουμε εδώ τον Επίτροπο, χαιρετίζω και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, Γενικού Διευθυντή, ο οποίος παραμένει ε, με το πουκάμισο, χωρίς σακάκι, αλλά σε εφέτος, ιδιαίτερος εφέτος, η Επιτροπή διαδραμάτισε με τρόπο επικοδομητικό με πνεύμα συνεργασίας τον ρόλο του α, καλού διαμεσολαβητή όπως της αρμόζει, ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά. Και ξέρουμε ότι πολλές φορές μας συμβαίνει να ε, καταφερόμεθα με σκληρά λόγια κατά τον εκπρόσωπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τώρα ήρθε η ώρα να τους ευχαριστήσουμε όλους. Merci. Alors, bien entendu, nous n'en resterons pas Βεβαίω δεν θα περιοριστούμε μόνο στα λόγια, όπω επιβάλλει η παράδοση. αμέσω μετά την ψηφοφορία του προπολογισμού την Τετάρτη, η ομάδα η πολιτική ομάδα του συντονιστή που έχει επιληφθεί μας προσκαλεί για ένα ποτήρι σαμπάνια για να πανηγυρίσουμε τα αποτελέσματα εάν αυτά είναι θετικά της ψηφοφορίας. Κύριε Προσκεκλημένοι, όλοι εδώ παρόντες, όσοι έχουν εργαστεί για αυτή την υπόθεση, ευχαριστώ πολύ την Άν για την πρόσκληση αυτή, την οποία απλώς μεταφέρω εκ μέρους της αλλά βεβαίω και τη δέχομαι εφόσον ε, είμαι και εγώ προσκεκλημένο. Αλλά για να μην φύγετε αμέσω, έχω να πω ότι έχουμε το σημείο 13 και το σημείο 14. Με δύο εκθέσεις κυρίες Καρβάλιο, η θέσπιση προγράμματος επιτήρησης και υποστήριξης. Με τρεις ή τέσσερις τροπολογίες, κύριε Καρβάλιο, υποστήριξη για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματο. Έχετε. Οι Κορσικανοί ναι, και οι Πορτογάλοι βλέπω αντιδρούν. Λοιπόν, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Ουδής. Ομόφωνα λοιπόν, χωρίς αποχές. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Ο κύριος Χάρτον. Καλά. Αποχές. Γκρίνεται. πέντε υπέρ. Κατά. Ε, αυτό θα συνοχλεί βέβαια. Μία, δύο, τρεις αποχές. Εγκρίνεται, να με άλλες αναλογίες. Καρβάλιο υπαριθμών 6 με προφορική τροπολογία. The Union, η Ένωση, η Συμβολή της Ένωσης και όχι η μέγιστη συμβουλή. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Τρεις. Και ένα μπιμπιπ που ακούστηκε στο μικρόφωνο. Τα, τα θα σημειώσουμε παρόλα αυτά. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχουμε τις πληροφορίες. Επτά. Τη συγκητρία υπέρ κατά. τρεις εποχές εγκρίνεται. Και ρωτώ αν μπορώ την 8, 9, 10, 11, όχι, δεν καταπίπτει. Θα κατέπεπτε αν είχε απορριφθεί 7. 11, 12, 11 μάλλον. 8, 9, 10 μόνο. Καλά, άντε, 8, 9 μόνο. Υπέρ. Κατά. Κατά, καλά, δηλαδή καταψηφίστε, αποχές, ωραία, οι 8 και 9 εγκρίνονται. 10, 11 μαζί, όχι, 10. Κατά, Αποχέ. εγκρίνεται 12, 11 υπέρ. Κατά, αποχές. Με μία αποχή εγκρίνεται. 12. Μα την, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 μήνα υπέρ. Συγκεκριμένη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ετυλογικές σκέψεις. Ε, μία της κυρίας Καρβάλιου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 μήναρ, συμβατή η συγκίτρινη υπέρ υπέρ, κατά. Αποχές συγκρίνεται 2. Καρβάλιο. Τεχνική φύση δεν Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. 31 υπέρ. Μία ψήφος κατά. Τρεις εποχές και συγχαρητήρια κύριε Καβάλιο. Και να δούμε αμέσως και το δεύτερο πρόγραμμα, τη δεύτερη έκθεση. Πρόγραμμα Κοπέρνικος. Και βλέπουμε τις 6 και 7 μαζί. Α συντονιστούν λίγο οι 6 υπέρ. Κατά. Μία ψήφο κατά. Αποχέ ε, εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. 1, 2, 3. Αποχέ εγκρίνεται. Η 7 κατά πίπτη. Η 22 κατά πίπτη. Η 8. Καταπίκτη. Όχι, έχει απορριφθεί. Έχει εγκριθεί 7, λέει ο μιλητή. 8, 9, 10, 11 μαζί. Ναι, ωραία. 8, 9, 10 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 του κυρίου Μινάρη, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 12 καρβάλιο υπέρ. Κατά. Αποχές μία. Απορρίφθη. Εγκρίνεται διορθώνει ο μιλητής. Με συγχωρείτε. Συμφωνείτε ότι εγκρίνεται, έτσι. Ωραία. Με όρασή μου. Την 23 του κυρίου Μινάς υπέρ, Κατά, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Παρά τις κάποιες παραστρατημένες οριστικές ψήφους. Η 13 Καρβαλιό. 25. 25 το κύριο ρίσει και υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Α, μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις ε, υπόλοιπες προτάσεις. Ψηφίζουμε τη 13 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ομού της 14, 15 και 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται, 17 υπέρ, κατά, με μία ψήφο, κατά, αποχές εγκρίνεται, 18 Βέρτμαν, η είναι κατά υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Μία και δύο τις συλλογικές υπαριθμών ένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η δεύτερη υπέρ. Κατά. Τρεις. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίσουμε την τρία. Την τέσσερα τώρα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται ομόφωνα. 19 Βέρτμαν. Συμβατή. Η υπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα. 20 του κυρίου Μινάρ. Αντικαθιστά τη λέξη ubiquity από το omnipresence, πανταχού παρουσία. Έχει μεγάλη διαφορά, ξέρετε, το ένα από το άλλο. μεγάλη λογοτεχνία, υπέρ, κατά, αποχές. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι οι δύο πολιτικές ομάδες προτιμούν το ubiquity από το omnipresence. Και όταν εξηγήσετε στους ψηφοφόρους σας αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα εκφράσω τον αμέριστο θαυμασμό μου, γιατί έχουμε φτάσει σε δυσθεώρατα φιλοσοφικά ύψη εδώ. Τέλο πάντων, ξεφεύγουμε από τα πεζά του προπολογισμού. Ε, στη συνέχεια του κυρίου Μινάρ, η συγκεντρία είναι κατά. Υπέρ, όχι, απε, ε, καταπίπτει γιατί 23 έχει απορριφθεί. Πάμε στην 5. Υπαριθμόν 5 πρέπει να ψηφιστεί. Υπέρ. Κατά. Άποχες Ενεκρίθη. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ, πέρα της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή και συγχαρητήρια κυρία Καρβάλιο. Μπορούμε λοιπόν τώρα ε, συνεχίζουμε με το 15. Είναι η έκθεση του κυρίου Νταρντέν, ο οποίος παρευρίσκεται. λοιπόν, έχετε όλοι το κατάλογο ψηφοφορία τη έκθεση Νταρντέν. Η ικανότητα των κρατών μελών τη Ένωση να αρχίσουν εγκαίρω και με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα τη νέα περίοδο προγραμματισμού τη πολιτική για τη συνοχή. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες του κυρίου Κοσλόφσκι και θα επιθυμούσα να τις ψηφίσουμε ομού. Διαφωνεί κάποιος επίμονο. Ωραία. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Γκρέτε. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης. Η πέντε ήταν ταυτόση με την τέσσερα. Η έξι έχει αποσυρθεί. Ωραία τροπολογία είναι αυτή. Επτά. Και επτά αποσύρεται λέει ο κύριος Μόλτερ. Ευχαριστώ Γιάν. Ορίστε άμα θέλετε. Οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η εννέα προφορική τροπολογία του εισηγητού απλούστερες διαδικασίες ζητεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στη τελική ηλεκτρονική πλέον ψηφοφορία Πέρασε. Αν ψηφίσατε όλοι. 27 υπέρ, 3 ε, κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Νταρντέν. Και τώρα ακολουθούν τα αγαπημένα μας θέματα. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, κύριε Σεγητά, μ' ακούτε, παρακαλώ προσοχή εδώ. Λοιπόν, μου λέγουν οι νομομαθείς μας ότι η τροπολογία σας υπαριθμών 1 ε, είναι απαράδεκτη νομικός πώς. Α, είναι και της δικής μου πολιτικής ομάδα. Απευθύνομαι λοιπόν στην πολιτική μου ομάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά τις προσπάθειές μου η ερμηνεία που δίνουν οι νομικές υπηρεσίες είναι ότι είναι απαράδεκτη η τροπολογία μας. Λυπούμε πάρα πολύ. Δεν θα τη θέσω σε ψήφιση, αλλά ε, το επιζητούμενο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί αν ψηφίσουμε το τελικό πρωτόκολλο. Οπότε είμαστε εντάξει. Δηλαδή, όσοι υπερψηφίζουν απορρίπτουν το πρωτόκολλο. Έτσι δεν είναι, γιατί αυτή είναι ε, η έκθεση του κ. Αλφόνση στο συμπέρασμά του απορρίπτει το πρωτόκολλο. Όποιος καταψηφίζει την πρόταση ε, και τα συμπεράσματα του εισηγητού ε, υπερψηφίζει, υιοθετεί το πρωτόκολλο. Εντάξει. Αμέσως λοιπόν και ηλεκτρονικός τελική ψηφοφορία. Τα καταλάβατε έτσι. Το ναι είναι όχι και το όχι είναι ναι. Εγώ τώρα τι να κάνω μέσα σε όλα αυτά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 9 ε, υπέρ, 23 κατά 0 αποχές. Άρα το πρωτόκολλο εγκρίνεται. Απορρίπτονται τα συμπεράσματα του εισηγητού. Πολύ ωραία, λαμπρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, αυτό ήταν για το Μαρόκο, ξέχασα να σας πω. Ε, γιατί οι μεγάλες περιπέτειες του Φρανσουά Αλφονσί δεν τελειώνουν στο Μαρόκο, γιατί συνεχίζει και μας προτείνει επίσης να προτείνουμε για ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με τη δημοκρατία της Γκαμπών. Ε, τώρα είναι υπέρ. Ε, μία ψηφοφορία λοιπόν υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται ωραία πάει και το καμπόν και οι δύο εκθέσεις για την Αλία. Τώρα έχουμε μια έκθεση του Τζοβάνι Λαβία για τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν αφενός τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και αφετέρου την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Βασικά όλη τη διατροφική αλυσίδα αφορά αυτό, την υγεία ε, ανθρώπων, ζώων και φυτών. Συν γυναικόπαιδα, ανάπηροι, χείρις, ορφανά κτλ. Τέσσερις τροπολογίες έχουμε εδώ του εισηγητού. Άλλα μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Φανταστικά. Υπέ Κατά. Ένας. Κατά άποχες. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά πάντα, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα και χρειάζεται οπωσδήποτε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Ένας αποκοιμήθηκε. 30 υπέρ, ένας κατά μία αποχή, συγχαρητήρια κύριε Σιγητά μας. Η απουσία του βέβαια. Bien, alors. Ωραία. Ε, λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε μεταφορές πιστώσεων. Σας παρακαλώ μην αποχωρείτε και μην ε, συζητάτε. Έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. Έτσι, η μεταφοράς απουσιάζει ο εισηγητής. Ε, είναι μία μόνη αίτηση μεταφοράς, παριθμόν 30 που αφορά ε, την ανάληψη υποχρεώσεων 5 εκατομμύρια χρειάζονται εδώ για τα μέτρα παρέμβασης ε, για αγορά ηχθείων για το 2013. Ε, υπάρχει αλλαγή στην νομική βάση. Στην Κόμπου News έχετε τις λεπτομέρειες. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Ο Ντέρεκ Βον βρίσκεται, θα μας πει για τα άλλα τμήματα. Μπορείτε να τα παρουσιάσετε unblock, Ντέρεκ, για όλα τα όργανα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καθώς τελειώνει η χρονιά, προφανώς ε, ε, τα αιτήματα για τις μεταφορές πιστώσεων αυξάνονται. Γι' αυτό έχουμε και από την Επιτροπή Περιφερειών και ε, τέσσερις μάλιστα, το διαμεσολαβητή, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Ελεκτικό Συνέδριο. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Κόμπου News που το έχετε φαντάζομαι στα χέρια σας για να διαβάσετε και τις λεπτομέρειες. Υπάρχει και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ένα αίτημα για μια μικρή μεταφορά. Μικροποσά είναι, εκτός από δύο και επειδή είναι ε, μεταφορές πιστώσεων είναι και δημοσιονομικά ουδέτερες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και συνιστώ στους συναδέλφους να δεχτούμε όλα αυτά τα αιτήματα για μεταφορά πιστώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Donc, si je comprends... Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, αν κατάλαβα καλά. Οι τέσσερις πρώτες ε, μεταφορές είναι προς ενημέρωση. Όχι, όχι. Νομίζω πρέπει να τις ψηφίσουμε και αυτές. Αμπλοκ όμως, μαζί. Ωραία. Ψηφίζουμε τις τέσσερις ε, μεταφορές πιστώσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τώρα, για το διαμεσολαβητή. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Υπηρεσία εξωτερικής δράσης, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το ελεγκτικό συνέδριο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει και άλλη μεταφορά πιστώσεων από την ε, ε, ΟΚΕ, η οποία όμως διατίθεται ε, μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας. Δεν τη γράφει το κόμπου News. Μπορούμε να την ψηφίσουμε τώρα ή την επόμενη φορά. Ο εισηγητή είναι υπέρ, δεν υπάρχει καμία ένσταση και για να κερδίσουμε χρόνο προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Κτηριακή πολιτική δεν έχουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Θαυμάσια. Θα παραχωρήσω την Προεδρία στον Ζαν Λουκντάν και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ah,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 Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε ακριβώ τώρα. Ε, το επόμενο θέμα λοιπόν με την λεγόμενη κινητοποίηση του EGF. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Έχουμε ήδη πει ότι υπάρχει μια ομάδα ε, η οποία ε, έχει απολυθεί από μια μεγάλη εταιρεία η οποία κατασκευάζει ε, μονάδες παραγωγής ρεύματος από αιωλική ενέργεια. Ζητούνται να ληφθούν μέτρα λοιπόν επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης, επανακατάρτισης και στήριξη σε αυτών που θέλουν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό είναι μια ιδέα η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προτείνει να δοθούν 6.364.000 ευρώ. Ζητείτε λοιπόν να εγκριθεί η μεταφορά. Έχουμε ήδη το 25% ε, προσημειωμένο θα έλεγε κανείς για την συγκεκριμένη αυτή χρήση. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο που διαφωνεί. Το επόμενο θέμα Ταμείο Παγκοσμιοποίησης 9,8 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε 4.000 απολυμμένους της επιχείρησης Nokia στη, μετά το κλείσιμο της μονάδας της. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ε, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και υπάρχουν αρκετά. Υπάρχει όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα θα έλεγα υποδειγματικού, παραδειγματικού χαρακτήρα επιχείρηση εμβληματική για την Ευρώπη στις νέες τεχνολογίες η εταιρεία Nokia. Νομίζω ότι το βασικό εδώ είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Η Φιλανδία έχει ε, μία βέβαια από, τις χαμηλότερες, ε, από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας. Είναι η τέταρτη φορά που κινητοποιείται το συγκεκριμένο ταμείο για την επιχείρηση αυτή, δύο φορές στη Φιλανδία, μία φορά στη Γερμανία και μία στην Ρουμανία συνολικά ε, έχουν πάρει 24 εκατομμύρια για 7.500 εργαζομένους. Η Νόκια απασχολούσε ε, στην Ευρώπη έναν στους πέντε εργαζομένους στην υψηλή τεχνολογία και είναι παρούσα η επιχείρηση αυτή σε σημαντικές επιχειρήσεις όπως η Ινδία και η Κίνα. Ε, απασχολούσε 60.000 ε, εργαζομένους, έχει όμως χάσει 10.000 και κάτι εργαζομένους. Η συναρμολόγηση των κινητών τηλεφώνων που γινόταν σε αυτά τα εργοστάσια μετακινήθηκε στην Κίνα, στην Νότια Κορέα, στην Ινδία και στο Βιετνάμ γιατί έτσι μπορεί κανείς συνεργαζόμενος με υπεργολάβους να προχωρήσει και να γίνει πιο ανταγωνιστικό σε επίπεδο τεχνολογίας. Το πακέτο χρηματοδοτείται κατά 50% από την φιλανδική κυβέρνηση. Υπάρχουν υπηρεσίες για την στήριξη νέων εργοδοτών έτσι ώστε να ξεκινήσουν τις δικές τους μορφές απασχόλησης. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη από το 2007 έχουν βοηθηθεί ε, από το Ταμείο αυτό 100.000 ε, εργαζόμενοι με ένα ποσό που φτάνει περίπου το μισό δις. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα και μια γεωγραφική ισορροπία. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο επιτρέπει σε επίπεδο αρκετά χαμηλό να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εγκρίνουμε την κινητοποίηση του συγκεκριμένου ε, ταμείου. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Και η τελευταία χρήση του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ να υποστηρίξετε το αίτημα των γερμανικών αρχών για την βοήθεια από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από απολύσεις ε, σε εταιρείε ε, που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια ε, σύμφωνα πάντα με το άρθρο 68 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου του 1996 και του κανονισμού 987 του 2006 για τη δημιουργία και χρήση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Η εταιρεία αυτή είναι μια εταιρεία η οποία προωθεί την χρήση της, ελληνικής, ε, της ηλιακής ενέργειας. Οι απολύσεις ε, προκλήθηκαν από διαφορετικές αλλαγές στην αγορά. Η Κίνα δημιούργησε μια τεράστια θα έλεγα παραγωγή, ταυτόχρονα μειώθηκε η ζήτηση και αυτό οδήγησε στην πτώση των τιμών κατά 40%. Από το 2005 μέχρι το 2011 το ποσοστό των κινέζικων επιχειρήσεων αυξήθηκε από το 11% στο 45% και το γερμανικό ποσοστό έπεσε από το 64% στο 20%. Η πτώχευση της εταιρείας οδήγησε στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους και οδήγησε στην αύξηση στην περιοχή του Βραδεμβούργου της ανεργίας κατά 4%. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία υποφέρει από ανεργία 11,3% αν συγκρίνουμε με τον εθνικό μέσο όρο 7,4%. Ο προϋπολογισμός που ζητείτε είναι 4,6 εκατομμύρια. Το 50% δηλαδή 2,3 εκατομμύρια ε, θα προέλθουν από το Ταμείο της, ε, ε, για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. 475 εργαζόμενοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα για την επανένταξή τους στην αγορά απασχόλησης. Κατάρτιση, έρευνα, επιδόματα ανεργίας κτλ. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να εγκρίνετε την πρόταση για τη χρήση του συγκεκριμένου ποσού από το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα, ε, μακροπρόθεσμα ε, Ευρωπαϊκά Ταμεία Επενδύσεων. ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη στην παρουσία της νομοδότησης αυτής είναι το γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων σε σχέση με το νέο κανονισμό που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επενδυτικά ταμεία και μακροπρόθεσμες δράσεις. Τι μπορούμε να πούμε εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμού. Με ικανοποίηση δεχόμαστε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αν θυμάστε καλά, στην προηγούμενη έκθεση για τα χρηματοοικονομικά μέσα ήταν από τα μείζωνα αιτήματα που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φέρει ένα κανονισμό Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή για να μπορέσουμε να συνενώσουμε όλους τους κανονισμούς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουμε νομική βάση επιτέλους ε, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν ε, μια ασφάλεια δικαίου και να μπορέσουν να ενοποιηθούν αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια μακροπρόθεσμα. Είναι γεγονός ότι η δική μας νομοδότηση δεν έχει μεγάλη ε, επιρροή, πώς να το πω, γιατί θα υπάρξει ένας οργανισμός εποπτικός που θα παρακολουθεί ε, αυτές τις δραστηριότητες, αλλά ε, θεωρήσαμε σημαντικό να γνωμοδοτήσουμε ακριβώς επειδή ήμασταν από τους εμπνευστές αυτού του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν καταθέσει και εννιά τροπολογίες, ορισμένες στις αιτιολογικές σκέψεις και άλλες στα άρθρα και ζητούμε καταρχάς βεβαίως και προφανώς η ΕΣΜΑ που θα είναι η αρμόδια αρχή να χειρίζεται αυτό το θέμα, να έχει τους απαραίτητους πόρους. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αρέσκεται πάρα πολύ στο να δίνει νέες ε, αρμοδιότητες στους οργανισμούς, αλλά δεν το συνοδεύουμε και με τους απαραίτητους πόρους για να απεξέρχονται σε αυτό το έργο. Επίσης, αν κάνουμε μια τροπολογία για να αυξηθεί, αν γίνεται, ο έλεγχος αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμα. Και δεν θέλουμε να συμμετέχουν χώρες που μπορούν να θεωρηθούν φορολογική παράδειση κτλ και να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου για αυτά τα ταμεία. Και σε ό,τι αφορά τα χρήματα οικονομικά μέσα, εάν κάποια στιγμή μέσω το χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης αν κληθεί να συμμετέχει ένα τέτοιο ταμείο, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Εν πάση περιπτώσει, καλωσορίζουμε την πρόταση. Εμεί συζητήσαμε και στο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα εγκρίνουμε την άλλη εβδομάδα προφανώ δεν θα λύσουμε τα προβλήματα των μεγάλων υποδομών που χρειάζονται μεγάλε επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα καλό τρόπο να κινητοποιηθούν όλε αυτέ οι αποταμιεύσει που περιμένουν να αξιοποιηθούν με τα απαραίτητα μέσα για να είναι ελκυστικό να συμμετέχει κανείς σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πολύ σύντομα. Δεν θέλω να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι το θέμα δεδομένων των αναγκών που έχουμε στην Ευρώπη για μάκρυ πρόθεσμες ε, ε, επενδύσεις αλλά και γιατί υπάρχει μια σημαντική βάση η οποία να είστε ακριβώς ε, μεσοπρόθεσμη απόδο, απόδοση στην επένδυση. Αλλά βλέπω δυστυχώς ότι κάποιες ε, από τις ε, παρατηρήσεις, κάποια από τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται, δεν αναπτύσσονται επαρκώς. Ενώ θα μπορούσε να είναι ένα πολύ δεδομένο προϊόν, το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι μόνο περιφερειακή σημασία. Σε σχέση με άλλα υφιστάμενα ταμεία είτε πρόκειται για τα ταμεία που γνωρίζουμε στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για ε, προϊόντα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, η δυνατότητα για δημοσιονομικές διατάξεις στα κράτη-μέλη, διαφορολογικές διατάξεις στα κράτη-μέλη, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη και ιδιαίτερα όταν μιλούμε για διάφορα νέα μέσα. Αναφέρθηκε δε, αλλά όχι επαρκώς, ότι τα παράγωγα προϊόντα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα πρέπει να προσαρμοστούν πολύ προσεκτικά σε αυτού τύπου στα μέσα, αλλά βλέπω εγώ ότι λείπουν κάποιες διευκρινήσεις όπως υπόθηκε νωρίτερα, ένα πολύ ενδιαφέρον μέσο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίτερα για τις υποδομές που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Με ένα μικρό σχόλιο μόνο, διότι συμφωνώ απολύτως με τη θέση του κυρίου Ρικέ. Ε, υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί καθόλου και έχω και κάποιες επιφυλάξεις. Όταν μιλούν για απόδοση των επενδύσεων πριν τη λήξη της επένδυσης. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα ε, το θέτει προς αξιολόγηση. Αλλά εμείς στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών δεν είμαστε αρμόδιοι για να κάνουμε όλες αυτές τις τροποποίησεις. Μήπως να τις υποβάλουμε απευθείας στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί εκεί είναι αρμόδια επί της ουσίας. Εμείς θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στη δημοσιονομική γνωμοδότηση. Και μάλιστα διευρυμένη την έχω ε, θεωρήσει σε αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα πραγματικά που δεν είναι καθόλου σαφή. Okay, thank you. Καλώς και ευχαριστώ. Έχετε τίποτα να πείτε εσείς για τον τριμερή. Άιβαλο. Α, ναι, ναι. Δεν έχουμε και τόσο πολλά να πούμε βέβαια. Απλώς σα για τις εξελίξεις. Έγινε η πρώτη συνεδρία στο τριμερούς για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα τέσσερα πρώτα άρθρα, τα πιο διαφιλονικούμενα, αυτά που έχουν να κάνουν με τα επίπεδα και το την αναλογία της διανομής, τη με το Συμβούλιο, θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα και προ... ετοιμάζουμε και συμβαστικές προτάσεις για τα σημεία τα οποία ήδη έχουμε επεξεργαστεί. Κύριες, αισθήματα δεν βλέπω. Τι επόμενε εβδομάδε θα έχουμε ίσως μια καλύτερη εικόνα από πλευράς ε, του Συμβουλίου για τα σημεία στα οποία υπάρχουν δυσκολίε. Η Επιτροπή ακολουθεί, παρακολουθεί προσεκτικά τις συζητήσεις. Περιμένουμε να δούμε το Συμβούλιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το, η Δευτέρα με το προσοχή τριμερή. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στην παρουσίαση της μελέτης. Η κυρία Νεπικιώση, η θα αναλάβει την Προεδρία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι πολύ σύντομη στην παρουσίαση της μελέτης, ώστε να αφήσω πιο πολύ χρόνο για τους ερευνητές μας. Ξεκίνησε αυτή η μελέτη μετά την Αραβική Άνοιξη και την ενισχυμένη ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δέσμευσή της. Έτσι έχουμε να κάνουμε με τροφοδότηση των προπολογισμών των εμπλεκομένων κρατών που πρέπει να παρακολουθείτε πάντως ε, ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι ε, γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Και λαμβανωμένη υπόψη και τη ενισχυμένη θέση Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Λισαβόνα και τη αποτελεσματικότητα εξοπλίση των κονδυλίων αυτών, Θέλουμε να έχουμε σωστή χρήση αυτών των κονδύλων στον προπολογισμό και θέλουμε επίσης να δούμε αν έχει κάποιο αντίκτυπο στη δημοκρατία, την προογωγή της δημοκρατίας, τον περιορισμό της φτώχειας κτλ. Εδώ επικεντρωνόμαστε στη μελέτη στην Αλγερία, την Αίγυπτο και την Τινησία, που έχουν ήδη ε, εφαρμόσει συστήματα ε, μέτρα υποστήριξη του προπολογισμού και που μας επιτρέπουν έτσι, στην περίοδο αυτή να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση. Η δημοσιονομική υποστήριξη δεν είναι αποτελεσματικό μέσο, πιστεύω, για την προαγωγή της δημοκρατίας, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη που από πλευρά τη ενισχύει τον εκδημοκρατισμό. Και θα ήθελα επίσης να καλέσω την ομάδα των ερευνητών τώρα να κάνει την παρουσίαση του έργου της. Θα τους βλέπω εδώ, όχι, σας είδα. Παρακαλώ. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα κύρια συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις μας από τη μελέτη αυτή. Επιτρέψτε μας συστηθώ. Η κυρία Βίλεμς και ο υποφαινόμενος εργαζόμαστε στις κάτω χώρες του Ρότζερταμ σε ένα γραφείο ε, παροχής συμβουλών, consulting, όπως αναφέρθηκε ήδη ο τίτλος της ε, μελέτης μας είναι η αποτελεσματικότητα της ε, παρεχόμενης βοήθειας της χώρας της Νότιας Μεσογείου. Επισημάνθηκε επίση ότι επικεντρωνόμαστε στην ε, την Ισία, την Αλγερία και, και την Αίγυπτο. Ε, τέσσερα κύρια θέματα μας απασχολούν. Εάν ο προπολογισμό, η υποστήριξη, η οικονομική υποστήριξη προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλαξε λόγω της Αραβικής Άνοιξης στην Αίγυπτο, την Ισία και την Αλγερία. Δεύτερο, εάν τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρέασαν τη δημοσιονομική ε, υποστήριξη και τα σχετικά προγράμματα στις χώρες αυτές. Μια τρίτη ερώτηση αφορά τα προγράμματα παρακολούθησης των προγραμμάτων δημοσιονομικής ενίσχυσης και επίσης μακροπρόθεσμα, τεταρτή ερώτηση, τι μπορούμε να αναμένουμε ως προς τη δημοκρατία των βασιμοτών δικαιωμάτων, την ενσωμάτωση της διάστασης των δύο φύλων, τη μείωση της φτώχειας από αυτή την υποστήριξη. Αυτό το, αυτά τα τέσσερα σημεία στα οποία εστιάστηκε η, η μελέτη μας. Κάναμε τις σχετικές αναλύσεις και τρεις αποστολές από μια εβδομάδα κάθε μία για την κάθε χώρα, η Άνια και ο προφαινόμενος αναλάβαμε αυτές τις ε, επισκέψεις με υποστήριξη από τους ε, τοπικούς παράγοντες. Και επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε κάποιες ε, προκατακτικές παρατηρήσεις. Out of our chapter Ε, γιατί αφού επικεντρωθήκαμε στα ζητήματα που είχαμε ορίσει για την ε, μελέτη μας, θα να κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση των γεγονότων της Αραβικής Άνοιξης για τις τρεις αυτές χώρες και επίσης ενδεχομένως θα πρέπει να αναλύσουμε και να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στο τι εννοείται ως δημοκρατία. Προχωρήσαμε λοιπόν και στην ανάλυση της επάρκειας του προϋπολογισμού που στηρίζει τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είδαμε λοιπόν πώς εξελίχθηκαν οι δαπάνες αυτές και σε ποιο βαθμό η προώθηση της δημοκρατίας έγινε ε, ελήφθη υπόψη. Το τέταρτο θέμα ήταν μια ανάλυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας εξετάσαμε σε ποιο βαθμό η πρόθεση της δημοκρατίας αναπτύχθηκε στα πλαίσια του καινούριου, ε, ε, της καινούργιας συμφωνίας. Δεν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν μπορώ τώρα να σας αναφέρω όλα τα σημαντικά σημεία από το κεφάλαιο 2. Υπάρχουν όμως ορισμένα σημαντικά θέματα, αυτά τα οποία φαίνονται στη συγκεκριμένη διαφάνεια, Πρώτον, αναλύοντας την έννοια της δημοκρατίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η δημοκρατική μετάβαση απαιτεί χρόνο σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη και η εμπειρία στην Αίγυπτο δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι βελτίωσης αλλά και περίοδοι πραγματικά όπου τα πράγματα πηγαίνουν ανάποδα. Δεν υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια στις εξελίξεις απαιτείται χρόνος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει κανείς τους στόχους στα πλαίσια της διάρκειας μιας δημοσιονομικής παρέμβασης η οποία κρατάει ένα, δύο, το πολύ τρία χρόνια. Αυτή η διαδικασία λοιπόν απαιτεί στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι ε, μεγαλύτερο χρόνο. Ταυτόχρονα εμείς ε, εννοώ εκ, εκτός των συγκεκριμένων χωρών. Οι εξωτερικές δυνάμεις βέβαια παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν παίζουν αποφασιστικό ρόλο, είναι περιορισμένος ο ρόλος τους και αν θέλει κανείς να δει τις, ε, ιδιαίτερα σε σχέση με την επιρροή της δημοσιονομικής βοήθειας. Ε, φυσικά θα πρέπει να γίνει σεβαστή και η εθνική κυριαρχία των χωρών αυτών, η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Το θέμα της στήριξης της ε, δημοκρατίας εμπεριέχει φυσικά και το θέμα ε, σεβασμού της εθνικής τους κυριαρχίας. Τέλος, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η δημοσιονομική βοήθεια για την προώθηση της δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν. Ως προς το πολιτικό πλαίσιο, τα μέσα τώρα υποστήριξη τη υποστήριξη, ε, όταν προτάθηκαν από τι αρχέ του αιώνα και με τι κατευθυντήριε γραμμέ που δημοσιεύτηκαν το 2002, αρχικά δεν είχαν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη δημοκρατία, να έχουν κάποια πολιτική επιρροή. Είχαν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν ε, τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ε, για την καταπολέμηση τη φτώχεια και να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, και με αυτό το πνεύμα ε, αναπτύχθηκαν αυτά τα μέσα. Άρα δεν μπορούμε να θεωρούμε πως ε, είναι δεδομένο ότι τέτοιου είδους μέσα, σχεδιασμένα δηλαδή για άλλους στόχους, μπορούν να είναι χρήσιμα και για την προαγωγή της δημοκρατίας, όσο και να θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για το στόχο αυτό. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος πάντως ότι τα καταφέρουν. Και έτσι έρχομαι στο επόμενο θέμα, ότι πράγματα πρέπει να γίνεται σαφής ε, διάκριση μεταξύ της προαγωγής της δημοκρατίας ε, και μιας ε, ως προϋπόθεσης για την παροχή της βοήθειας και της παράπλευρης ε, συνέπειας αυτής της βοήθειας. Εδώ λοιπόν μέχρι το 2007, αν και θα πρέπει να πω μέχρι το 2012 πιο σωστά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη βοήθεια ορίζει δύο στόχους, τον περιορισμό της στόχιας και την υποστήριξη οικονομικής ανάπτυξης. Μόνο με τις πρόσθετες του 2012 ενσωματώνεται ένας νέος στόχος προαγωγή δηλαδή της δημοκρατίας. Στις 10 δευτερίες γραμμές για το 2012 βλέπουμε ότι είναι και στόχος αλλά και προϋπόθεση η προαγωγή της δημοκρατίας. Θα επανέλθω όμως αργότερα σε αυτό. Και επίσης θα πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ της γενικής ε, δημοσιονομικής ε, στήριξης και της ειδική, γιατί στην ε, γενική έχουμε ένα διάλογο σε μακροοικονομικό επίπεδο με την ε, χώρα που αποδέχεται αυτή την βοήθεια και κάνουν πιο γενικό συνδυασμό. στο πιο συγκεκριμένο όμως ε, διάλογο για τον προπολογισμό εστιαζόμαστε σε τομεακές πολιτικές με συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκουμε και προσπαθούμε να ε, υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν το να προσπαθήσουμε να σωματώσουμε πολιτικά αποτελέσματα στο επίπεδο αυτό ε, έχει μεγαλύτερο νόημα στον, ε, στην γενική δημοσιονομική υποστήριξη και όχι στην ε, τομεακή. Αυτά ως προς την εισαγωγική μας τοποθέτηση που έχει αναλυτικό χαρακτήρα μάλλον. Θα μπορούσα να πω και πολλά άλλα πράγματα, αλλά θα τα αφήσω προς το παρόν. Για δε την Αίγυπτο. που έχει θέματα για την εκπαίδευση, την δημόσια υγεία, την ίδρυυση, το περιβάλλον, τις μεταφορές, προγράμματα που χρηματοδοτούνται, προγράμματα που έχουν διατυπωθεί ήδη πριν από την Αραβική Άνοιξη, κανένα δύο χρόνια πριν την Αραβική Άνοιξη και που υποστηρίζουν τομεακές πολιτικές με στόχο την υλοποίηση κάποιων τομεακών ε, στόχων, στόχων που παραμένουν ε, ισχυροί, δεν έχουν δηλαδή ανατραπεί λόγω της Αραβικής Άνοιξης, δεν έχουν αναιρεθεί λόγω της Αραβικής Άνοιξης και γι' αυτό όπως θα διαπιστώσετε δεν έχουν αναδιατυπωθεί λόγω της Αραβικής Άνοιξης αυτές οι στοχεύσεις, ε, παραμένουν και υλοποιούνται. Το πιο σημαντικό ως εμπόδιο που διαπιστώνουμε στα θέματα αυτά είναι το ότι είναι πιο δύσκολη η πιστοποίηση μετά την Αραβική Άνοιξη λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε σε πεδίο ε, κρατικού μηχανισμού. Ε, δεν υπάρχουν σαφείς ε, κατευθυντήριες γραμμές, είναι πιο δύσκολη η υλοποίηση, αλλά ο στόχος, το περιεχόμενο, η περιγραφή των προγραμμάτων δεν έχει αλλάξει. Πέραν τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει συζητήσεις ε, με, τις με την κυβέρνηση της Αιγύπτου το 2012 για την ανάπτυξη μιας σύμβασης ε, συμφωνίας ε, οικοδόμηση κρατικού μηχανισμού που αποτελεί τη νέα μορφή συνεργασίας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι εδώ βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα περιλάβει η δημοσιονομική βοήθεια ε, προϋποθέσεις ε, στον στόχο του εκδημοκρατισμού αν και δεν μας έχουν αποκαλύψει τι είδους προϋποθέσεις θα είναι αυτές τουλάχιστον ε, στις διαπραγματεύσεις που γίνονταν μέχρι τον Απρίλιο εφέτος με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Πάντως είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να ξεκινήσει ούτε καν την υπογραφή πόσο δε μάλλον τη χορήγηση των ποσών, ε, εάν δεν έχουν φτάσει σε κάποια επίπεδα ικανοποιητικά οι Αιγύπτιοι και για τη μακροοικονομική ε, πολιτική και για την διαχείριση των κονδυλίων. Ε, μέχρι τη στιγμή που είχαμε μείνει ήταν πολύ περιορισμένες οι πρόοδοι και γινόταν μια προσπάθεια μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αφρική Τράπεζα Αναπτύξεως και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, θέλουμε να το περιλάβουμε και αυτό, δηλαδή σε, τέσσερα, σε πέντε τεσσάρων θεσμικών φορέων. Έτσι είχε η κατάσταση τότε. Έρχομαι τώρα στην Τινησία. Είναι διαφορετική η κατάσταση και από την Αίγυπτο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει ενίσχυση στην Τινησία ε, γενική του προπολογισμού ήδη από το 2008 αν δεν απατώμε. Και αυτή τη φορά ήταν περισσότερο εστιασμένη στην οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Τα ποσά δεν ήταν τεράστια, ήταν περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι σχετικά μικρό πόσο αν σκεφτεί κανείς την οικονομία της ε, Τινησίας, αλλά υπήρξαν και άλλοι δωρητές αρκετά γρήγορα μετά την Αραβική Άνοιξη, πότε ήταν αυτό το Μάρτιο δηλαδή, ε, τον Απρίλιο του 2011, άρχισαν οι δωρητές μια καινούργια συζήτηση με τη νέα κυβέρνηση για οικονομική αλλά και πολιτική υποστήριξη για ένα νέο ε, είδος ε, υποστήριξης γενικής του προϋπολογισμού και οι νέες συμβάσεις αφορούσαν την κοινωνική ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ε, καταπολέμηση κάποιων κοινωνικών προβλημάτων και κάλυψη κοινωνικών ε, αναγκών της κοινωνίας, που ήταν άλλωστε και ε, η υπόθεση που πυροδότησε την Αραβική Άνοιξη. Αυτά είναι από το γενικό βοήθημα για τον προϋπολογισμό. Στη συνέχεια το 2011 και το 2012, καθώς και το 2013 στις αρχές, πήγε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρχισε να συζητάει ένα νέο πλαίσιο για μια γενική ε, και πάλι σύμβαση για την οικοδόμηση του κράτους. Εμείς είχαμε πάει εκεί το Μάρτιο-Απρίλιο του 2013. Δεν υπήρχε ουσιαστική πρόοδος γιατί είχε επιδεινωθεί η πολιτική κατάσταση. Θυμάστε ότι στις εφημερίδες ε, αναφερόταν πολιτική αστάθεια, και γενικότεροι, οι τρεις δωρητές, δηλαδή η ε, Αφρικανική ε, Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρίτος δωρητής τήρησαν μια στάση αναμονής. Και, ε, υπήρχαν και δύο τομαϊκά προγράμματα για υποστήριξη προϋπολογισμού. Τι ήταν η ίδρυυση και το περιβάλλον, αν δεν απατώμε και για αυτούς τους τομείς ισχύουν τα ίδια με την Αίγυπτο. Είχαν αρχίσει συνεργασίες ε, νωρίτερα και ως στόχοι πριν την Αραβική ε, Άνοιξη και η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη και η τομεακή υποστήριξη και οι συμβάσεις γενικότερα. Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα λόγω της Αραβικής Άνοιξης. Έρχομαι τώρα στην Αλγερία και πάλι τελείως διαφορετική η κατάσταση διότι η Αλγερία είναι μια χώρα πλούσια σε ό,τι αφορά τους ε, δημοσιονομικούς πόρους έχουν πολύ ε, πετρέλαιο αλλά κυρίως ε, φυσικό αέριο που εξάγουν οπότε είναι σε μια άνετη δημοσιονομική θέση. Ο γενικός προϋπολογισμός ποτέ δεν υποστηρίχθηκε, ούτε το είχε σκεφτεί καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε άλλοι δωρητές, δεν είναι ζήτημα αυτό. Ένας τομέας που υποστηρίζουμε δημοσιονομικά συνεχίστηκε που ήταν για την ίδρυψη και το δεύτερο που προετοιμάζεται είναι για το περιβάλλον. Αυτά τα προγράμματα υποστήριξης ε, του προπολογισμού δεν εδόθησαν επειδή ε, χρειαζόταν χρήματα η κυβέρνηση, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να αλλάξει το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας και να εστιάσει σε τομείς πολιτικών, θεσμικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Και όταν κάνεις τέτοια προγράμματα και τέτοιου είδους συζητήσεις πρέπει να υπάρχει και μια στόχευση με τομεακή στήριξη του προπολογισμού, όχι με μονομένα προγράμματα. Έχω γράψει εδώ ότι δεν υπήρχε καμία επιρροή από την Αραβική Άνοιξη, είναι πολύ απόλυτο. Θα έλεγα μικρή επιρροή και πολιτικά και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βοήθειας. So, Αυτά είναι τα τρία κράτη που αναλύσαμε και ας δούμε τώρα τη μελέτη για να απαντήσουμε στα θέματα της πρώτης μελέτης. Έρχομαι στη δεύτερη μελέτη. Η μελέτη λοιπόν ασχολήθηκε με πέντε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάναμε λοιπόν ε, μία απογραφή και είδαμε πόσα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου αφορούσαν την ε, υποστήριξη του προπολογισμού. Δεν ήταν πάρα πολλά, αλλά δεν είχαμε πολλά πράγματα να αναφέρουμε. Είναι πέντε λεγότα τα ψηφίσματα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένα με την Αίγυπτο μετά το 2011. Ε, ένα ψήφισμα είχε σχέση και ήταν κάτι που αφορούσε τη μελέτη μας. υποστήριξη ε, του προπολογισμού θα πρέπει να διατηρείται ε, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτους δικαίου. Είναι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Ε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, από το 2011 έχει στείλει μια αντιπροσωπεία που εργάζεται ε, πάντα στα πλαίσια αυτού του ψηφίσματος. Διότι τι κάναμε ε, ως γενική υποστήριξη του προϋπολογισμού. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις, συμμετείχαν σε συζητήσεις, άρχισαν τις προετοιμασίες, αλλά δεν δεσμεύτηκαν πάρα πολύ γρήγορα με δεσμεύσεις απέναντι στη νέα Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήταν σωστή αυτή η προσέγγιση. Είδαμε και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την Τινησία και την Αλγερία, αλλά κανένα από αυτά δεν αφορούσε ε, θέματα δημοσιονομικά. Το τρίτο ερώτημα της μελέτης ήταν η παρακολούθηση και η αναφορά. Ε, τι είναι αυτό στα πλαίσια της στήριξης του προπολογισμού. Στην αρχή πρέπει κανείς να διαπιστώσει ότι με τέτοια δημοσιονομική βοήθεια που δεν είναι project, δεν είναι έργο, πολιτικές και δράσεις υποστηρίζονται ε, στις δικαιούχες χώρες ή στα Υπουργεία και εκείνοι κάνουν και την παρακολούθηση και την αναφορά. Αυτό το αναφέρει ρητά και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, της εκάστοτε κυβέρνησης. Λοιπόν, κοιτούμε τι έχουν κάνει εκεί. Τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Υπάρχουν μερικά υπουργεία που τα πηγαίνουν καλά και άλλα που έχουν λιγότερο καλές επιδόσεις και ακριβώς επειδή αποδυναμώθηκαν οι κυβερνήσεις το 2011-2012 και στις τρει χώρε ε, μειώθηκε και η ποιότητα μοιραία των αναφορών αυτών. Λοιπόν, άλλη παρατήρηση. Τι μας αναφέρουν κυρίως σε σχέση με τη χρηματοδότηση τη δική μας και τις ε, αποφάσεις που λαμβάνονται και το καθαρό αποτέλεσμα. Αλλά για τον αντίκτυπο και το ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν είναι πολύ καλή η ε, αναφορά. Πρέπει να βελτιωθεί πολύ να μάθουν πώς να αναφέρουν τέτοια ζητήματα σε ό,τι αφορά την τομεακή υποστήριξη επιμέρους πολιτικών δεν έχει αλλάξει το περιεχόμενο, άρα δεν έχουν αλλάξει και οι δείκτες μέχρι κάποιου βαθμού. Η Γενική Υποστήριξη Προπολογισμού στην Δινησία, να πω δύο λόγια γιατί διαφέρει από τις άλλες χώρες, ε, εκεί εστιάζεται στην παρακολούθηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, μακροοικονομική σταθερότητα και άλλα. Και οι μακροοικονομικές πολιτικές αλλά και οι πολιτικές. Ε, αυτόν εστιάζουμε και επίσης εκεί δεν άλλαξε τίποτα γιατί δεν άλλαξε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι δείκτες είναι οι ίδιοι. Ορισμένα λοιπόν από αυτά τα στοιχεία και οι δείκτες έχουν να κάνουν και με τον αντίκτυπο και τις επιδόσεις ε, που σας είπα, αλλά αυτά είναι θέματα μέσω μακροπρόθεσμα, δεν μπορείς από τη μια χρονιά στην άλλη να κρίνεις. Τέταρτη ερώτηση για τη μελέτη, που είναι ίσως και το πιο ακαθόδες και το πιο φιλόδοξο και δύσκολο ερώτημα, ήταν Ωραία. Πώς μπορεί να βοηθήσει αυτή η οικονομική βοήθεια για να προωθηθούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, ζητήματα φύλου και μείωση της φτώχειας. Η πρώτη παρατήρηση την οποία θα κάνουμε σε αυτή τη σύντομη μελέτη, γιατί πήγαμε μόνο μία εβδομάδα σε κάθε μία χώρα, ε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε πάρα πολλά στοιχεία. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ερώτηση η οποία πράγματι απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις επιπτώσεις στη μείωση της ένδυας, αυτό είναι ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο στοιχείο και πρέπει να ακολουθήσει κανείς μια συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί και ο ΣΑΣΑΝ παράδειγμα ε, και απαιτείται ένας χρόνος περίπου για να ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή και κοστίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε μία πρωτότυπη δική μας ανάλυση αποτελεσματική. Μπορέσαμε όμως να κάνουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις ε, για την τομεακή στήριξη του προϋπολογισμού. Σαν παράδειγμα παρεμβάσεις στον τομέα του καθαρού νερού, ε, της υγείας και της εκπαίδευσης. Ε, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα του περιβάλλοντος, συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορούν να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και να συνεισφέρουν έτσι έμεσα στη μείωση της φτώχειας. Για την προώθηση τώρα και τη στήριξη της δημοκρατίας, όπως σας είπα, ε, έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική η άμεση δημοσιονομική στήριξη για την προώθηση της δημοκρατίας. Υπάρχουν βέβαια έμεσες μορφές στήριξης. Μέσω της στήριξης του προϋπολογισμού μπορεί κανείς να προωθήσει την εμπλοκή του πληθυσμού, ε, να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τον πληθυσμό στον τομέα της υγείας, της παροχής νερού κτλ και του ελέγχου ακριβώς του δημοκρατικού των δημοσίων υπηρεσιών, κάτι το οποίο αυξάνει τη δημοκρατία, αλλά αυτά είναι έμεσες επιπτώσεις και όχι άμεσες για την πρόθεσή της. Λοιπόν, θα καθυστερήσω λίγο. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για τις συστάσεις τις οποίες θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε ε, στο τέλος ε, της παρουσίασής μας. Πρόκειται για τη σελίδα 48 του εγγράφου το οποίο σας έχει διανεμηθεί. Στην παράγραφο 5,2 παρουσιάζουμε πέντε συστάσεις. Η πρώτη σύσταση στο έγγραφό σας είναι η σελίδα 54. στη σελίδα 56 διορθώνει ο μιλητής. Υπάρχουν λοιπόν πέντε συστάσεις. Η πρώτη σύσταση συνδέεται με τις αμφιβολίες για την καταλληλότητα του μέσου δημοσιονομικής στήριξης για την προώθηση της δημοκρατίας. Δεν έχει, δεν έχει καταλήξει, δεν έχουμε και εμείς καταλήξει. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημοσιονομική στήριξη όμως, και θέλουμε εμείς να προωθήσουμε τη δημοκρατία και μέσω του προϋπολογισμού, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε καλύτερα τις δραστηριότητες και τις προϋποθέσεις που μπορεί να θέσει κανείς έτσι ώστε να καταστήσει την παρέμβασή του αποτελεσματική. Στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχουν και πολλές κατευθύνσεις. Λέγεται ότι είναι ένας στόχος, αλλά τίθεται το θέμα του πώς θα πετύχουμε τον στόχο αυτό. Πρώτη σύσταση. Δεύτερη σύσταση αναφέρεται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τα έγγραφα που τη στηρίζουν. Ε, η φράση ε, δεν χρησιμοποιείται στήριξη του προϋπολογισμού, έστω μία φορά ίσως και μόνο. Ε, υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως στο Κοινοβούλιο ότι η προαπόφηση της δημοκρατίας είναι ένας βασικός στόχος της πολιτικής γειτονίας. Η τρίτη σύσταση αναφέρεται στην ευαισθησία ε, της δημοσιονομικής στήριξης στις πολιτικές αλλαγές στις χώρες αποδέκτες. Η στήριξη του προϋπολογισμού είναι κάτι το οποίο σαν μέσο πολιτικά παρουσιάζει πάρα πολλές ευαισθησίες στις ευνίδιες αλλαγές στις χώρες που αποδέχονται τη βοήθεια αυτή. Αυτό σημαίνει ότι σε πολιτικά ασταθείς χώρες οι δωρητές θα πρέπει να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Η τέταρτη σύσταση Καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα για τις πολιτικές επιπτώσεις ε, της στήριξης της δημοσιονομικής. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στη γενική δημοσιονομική στήριξη και στις επιμέρους τομεακές στήριξης. Ε, πολλές φορές οι τομεακές στήριξεις είναι πιο αποτελεσματικές και πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα στις ασταθείς χώρες, ε, μπορεί να δοθεί μια τέτοια βοήθεια, ενώ δεν μπορεί να σταθεί, αν θέλετε, μια γενικά, ε, γενικής φύσεως χονδρική δημοσιονομική βοήθεια. Τώρα, στο τέλος, η τελευταία σύσταση αφορά την παρακολούθηση των εξελίξεων και της αποτελεσματικότητας της βοήθειας της κοινοτικής σε αυτές τις χώρες. Όχι μόνο επιδόσεις, αλλά κυρίως σε σχέση με τις πραγματικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank very much. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστώ την ομάδα των ερευνητών για τη δουλειά της. Η μελέτη αυτή ελπίζουμε ότι θα δώσει κανές πληροφορίες για το μέλλον της ε, ε, χορήγησης αυτής της βοήθειας ε, προς όφελος του Κοινοβουλίου. Η μελέτη αναλύει τον, τρόπο, τον βαθμό στον οποίο η δημοσιονομική υποστήριξη προσφέρεται έχει αλλάξει σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη και σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει στις δημοκρατικές με τα εξελίξει χώρε αυτέ. Πιστεύω ότι η μελέτη δεν έδωσε απαντήσει σαφεί σε όλα αυτά τα ερωτήματα ναι. και γι' αυτό θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Αν και δυστυχώ δεν έχει μείνει πολλή ε, κόσμο, εγώ τουλάχιστον έχω παρόντα συνάδελφο, πρώην υπουργό μάλιστα, των εξωτερικών, ο οποίο θα μπορούσε και να λάβει το λόγο εάν το επιθυμεί. Ερωτώ λοιπόν, θε να πει κάτι για τη μελέτη. Όχι, γιατί μπορούμε έτσι να κάνουμε κάποια σύντομα σχόλια για τα όσα μας παρουσιάστηκαν. Ναι, ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και είχα την ευκαιρία να ρίξω μια ματιά ομολογώ και εγώ, μας έχει απασχολήσει στο Κοινοβούλιο τι είδους τύπο και αποτελεσματικότητα μπορεί να προσλάβει αυτή η βοήθεια και αυτό και από πλευρά τη Επιτροπής ε, του Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει να σας πω ότι είναι το σημείο στο οποίο χωλένουμε ότι δεν βλέπουμε αποτελεσματικότητα. Και είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε για τη Βόρεια Αφρική, για τη Νότια Όφη της Μεσογείου. Γιατί έχουμε αρκετά αντιφατικά στοιχεία που προκύπτουν από τις μελέτες μας, από τις ερευνές μας, στην, κυρίως για την Αίγυπτο. Mm. Η... Μελέτη βέβαια το καλύπτει ένα βαθμό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η δημοσιονομική ενίσχυση είναι βέβαια κάτι το καλό. Τώρα το τι αποτέλεσματα συγκεκριμένα θα προσφέρει εκ των υστέρων. Τι αντίκρισμα συγκεκριμένα για τα κράτη-μέλη ή τι εναλλακτική ενδεχομένως θα υπήρχε με την χρηματοδότηση και συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι κάτι το ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω και η καταγραφή αποτελεσμάτων, η αναφορά δηλαδή, αλλά και τα συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελέσματα έχουν σημασία. Και ειδικά όταν μιλάμε για δημοσιονομική ενίσχυση, καλό είναι να έχουμε ορατότητα ως προς τα αποτελέσματα, ε, την ε, ε, πρακτική εφαρμογή, τα ποσά που εισραίουν σε εθνικούς προϋπολογισμούς και το καθεξής. Τώρα συζητώντας την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έχει βέβαια μια συγκεκριμένη εντολή και έχουμε να κάνουμε με την πολιτική γειτονία, είμαστε μοιρασμένοι μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, αλλά ένα από τα καυτά ζητήματα που μας απασχολούν στις στήσεις μας με την τράπεζα και τα μέλη είναι κατά πόσον πρέπει να αλλάξουν τα τα ανώτατα επίπεδα γίνονται διάφορες προτάσεις να κοιτάξουμε πιο πολύ προς Ανατολάς και λιγότερο προς Δυσμάς και αυτό πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον να το εξετάσουμε. Το επιχείρημα βέβαια είναι ότι οι πολιτικές αλλαγές ε, θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να φέρουν καρπούς και μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ευρεία κλιμακός χρηματοδότηση χώρε Δεν ξέρω αν έχετε κάποια προτίμηση, κάποιε ιδέε. Χωρί μικρόφωνο ο αναλυτή. Α, μάλιστα. Το βρήκα. Ε, καταρχάς, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν είμαι βέβαιος εάν ε, μπορεί με τη δανειοδότηση να υποστηρίξει προπολογισμό. Όχι, όχι, δεν λειτουργεί έτσι λέει ο κύριος Κάλφιν, αλλά καμιά φορά ε, ε, υπάρχει ένα μείγμα δανείων με μακροοικονομική βοήθεια. Αλλά είναι και θέμα εντολής, αλλά η πολιτική ευθύνη καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησεων. Δηλαδή, δίνουν φτηνή χρηματοδότηση για στοχευμένες δράσεις, για συγκεκριμένους τομείς που ε, συνάδουν πάρα πολύ με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Η όλη ιδέα λοιπόν είναι να ευθυγραμμιστούν οι ε, ευρωπαϊκές πολιτικές με τη δυνατότητα της τράπεζας να χρηματοδοτεί συγκεκριμένα έργα. Δεν περνάει μέσα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά ε, καμιά φορά ακριβώς υπάρχει ένα τέτοιο χαρμάνι, ένα συνδυασμός, ακριβώς τα ίδια έργα. Μάλιστα. Και κλείνει το μικρόφωνο ο μιλήτης. Λοιπόν, ναι, όντως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δανειοδοτεί ε, ε, για συγκεκριμένες περιπτώσεις στα κράτη, αλλά είναι, υπάρχει και μια πολιτική χρειά, αν θέλετε, για την τράπεζα. είναι παραχωρήσεις ουσιαστικά και έχουν και μια πολιτική χρειά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητο αυτό από πολιτικής άποψη από τη μακροοικονομική βοήθεια. Από χρήματα δηλαδή που πηγαίνουν στον προπολογισμό της χώρας κανονικά. Ε, και η γενική υποστήριξη του προϋπολογισμού ε, χρεώνει ας πούμε στο δωρητή τις οποιασδήποτε δράσεις και παραλήψεις μιας κυβέρνησης. Ενώ η κλαδική βοήθεια, η τομεακή, πηγαίνει σε συγκεκριμένες δράσεις, πολλές φορές ε, και είναι τελείως εκτός του προπολογισμού και εκτός ελέγχου ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες φορές περνάει μένα από το γενικό προϋπολογισμό, ε, είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά υπάρχει ειδική προσημείωση για το πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Και θα σας έλεγα επίση ότι η πολιτική ευαισθησία εκεί της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ακόμα μικρότερη καμιά φορά ε, σε σχέση με την υποστήριξη έργων, γιατί τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι εμπορικά δάνεια που χορηγούνται για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς και δεν περνούν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού συνήθως. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι σε χώρες ασταθείς μπορεί κανείς να δίνει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χωρίς υποστήριξη του προϋπολογισμού ή και ακόμα και ε, ε, βοήθεια για έργα που υλοποιούν οι ε, δικαιούχοι Κυβερνήσει, κυβερνήσεις. Εγώ δεν είμαι ειδικό για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κάποιες σκέψεις μοιράζομαι μαζί σας. Και μια που μιλούμε και για την προβολή της ευρωπαϊκής βοήθειας σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν δύο στοιχεία προβολής εκεί να βάλουμε σημαία, αλλά αμέσως μετά βλέπεις και τα αποτελέσματα της υποστήριξης. Ε, όταν μιλάτε για ορατότητα, για προβολή, ε, αυτό που σας ενδιαφέρει κυρίως είναι τα αποτελέσματα. Η προβολή τι σημαίνει, ότι αυτό το έργο έγινε με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν μπορείς, γιατί είναι μέσω του προϋπολογισμού. Μπαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα στο γενικό και στις κλαδικές επιμέρους ε, δράσεις, αλλά τουλάχιστον στα επιμέρους μπορείς να πεις ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι και κάποια στοιχεία πολιτικής που έχουν συζητηθεί και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές ε, οι προϋποθέσεις, δημιουργούνται νέοι θεσμοί, γίνονται νέες κινήσεις, νέες δράσεις αναλαμβάνονται και νέες πολιτικές υλοποιούνται και γι' αυτό έχει συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί προβάλλεται αυτό και μπορεί κανείς να το αναγνωρίσει. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς αυτό το σχολείο, αυτό το κέντρο υγείας, αυτό το αποχετευτικό έργο ή το αρδευτικό το έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Δεν ξέρω. Ρωτήσατε τίποτα άλλο ειδικό ή θέλετε να ρωτήσετε. Thank you very much. Is there somebody... Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει. Να κάνει καμία ερώτηση για τη μελέτη ή τίποτα άλλο γενικότερο. Anybody from the assistance? Κανείς βοηθός ίσως? No, it seems that it's not the case. Όχι. Νομίζω ότι ήταν εκτενής η παρουσίασή σας και εξαντλητική, οπότε κάλυψε και όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Κάλφιν για τη συμπροματική του ερώτηση που μας βοήθησε να καλύψουμε ένα ευρύτερο φάσμα. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος των συναδέλφων ε, για ε, το ε, αργό της ώρας, την ώρα που σας καλέσαμε να παρουσιάσετε τη μελέτη. Αυτό επηρεάζει και την παρουσία των βουλευτών, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν την ευκαιρία να τη διαβάσουν και βεβαίως να βασίσουν ε, τη μελλοντική τους εργασία και στη δική σας μελέτη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκτιμώ την ε, συνεισφορά σας. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Καλή σας ε, επάνωδο.